Uh, Αγαπητοί συναδελφοί, έχουμε πάρα πολλή δουλειά σήμερα, οπότε ας αρχίσουμε στην ώρα μας, αν δεν σας πειράζει. Αρχίζουμε λοιπόν με την έγκριση της ημερησίας διάταξης. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις, εγκρίνεται. Έγκριση των πρακτικών της 25ης Ιουνίου και 25ης Σεπτεμβρίου. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, στα πρακτικά αυτά επίσης θεωρούνται εγκεκριμένα. Ανακοινώσεις του Πρόεδρου για το γλωσσικό καθεστώς. Έχουμε διερμηνία σε όλες τις γλώσσες εκτός από τα δανέζικα, τα κροατικά και τα γκέλικ. Έγκριση τώρα των συστάσεων των συντονιστών. Ο ορισμός εισηγητών, ο κύριος Ντάλτον από το ECR ορίστηκε εισηγητή για την πρόταση κανονισμού όσον αφορά την πρόληψη διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Αντικαθιστά την κυρία Χέλγα Στίβενς. Συμφωνεί η Επιτροπή με τη σύσταση αυτή. εγκρίνεται. Στη συνέχεια, κατεξοδότηση και εκτελεστικέ πράξεις. Εκτελεστική πράξη τη 28 Νοεμβρίου του 2018. Το Κοινοβούλιο έλαβε ε, εκτελεστική πρόταση οδηγίας όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές για την σήμανση των πυροβόλων όπλων και των εκείνων συστατικών τους υπό την οδηγία του Συμβουλίου 91-477 και τώρα η βασική πράξη της οδηγίας 2017-853 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Μαΐου 2017 τροποποιούν την οδηγία του Συμβουλίου 91-477 για τον έλεγχο, για την απόκτηση και την κατοχή ε, πυροβόλων όπλων. Εάν υπάρχουν ε, αντιρρήσεις, ενστάσεις, να ξέρετε ότι έχει ανακοινωθεί η παραλαβή της πράξης αυτής μέσω του newsletter της 30 Νοεμβρίου 2018 και ετέθη και εσωτερική προθεσμία με την ε, ημερομηνία 12 Δεκεμβρίου 2018 στις 12 Έχουμε και ψηφοφορία σήμερα, 5,5 με 7 κατά πάσα πιθανότητα. Να έχετε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες μαζί για την ψηφοφορία, παρακαλώ. Φαντάζομαι ότι θα έρθουν και άλλοι ευρωβουλευτές μέχρι τότε. Πάντως ευχαριστώ τους παρόντες, να το ξέρετε. Άλλη μια ανακοίνωση έχω. Είσαστε προσκεκλημένοι να συμμετάσχετε σε κοινοβουλευτικό διάλογο των εκκλησιών και οργανώσεων βάσει του άρθρου 17 με αφιτρίωνα την ε, Μαρή Μαγκίνες, την αντιπρόεδρό μας. 4 Δεκεμβρίου ανθρώπινα δικαιώματα και εκκλησίες, επιμερισμένη ευθύνη. Θα είναι και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η πρώτη αντιπρόεδρος. Αυτές οι προσκλήσεις λοιπόν που είχα να σας μεταφέρω. Και τώρα περνάμε στην ημερήσια διάταξη αυτή καθεαυτή. Σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης πρόκειται για την ε, εφαρμογή του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εισηγητής ο κύριος Ντανίς Τεγιόγκ μας παρουσίασε ε, το κείμενό του. Έχουμε 67 τροπολογίες, οπότε τώρα θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων για τις τροπολογίες αυτές. Οπότε παρακαλώ ο κύριος Ντεγιόγκ που είναι ο εισηγητής μας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος γιατί βλέπετε και πόσο πολύ είμαστε εδώ ε, γι' αυτό το τόσο δύσκολο και ενδιαφέροντα φάκελο. 67 τροπολογίες, ναι. Οι περισσότερες από αυτές βελτιώνουν το κείμενο και συστήνουν να τις υπερψηφίσουμε. Υπάρχουν και αυτές που θέλουν διαγραφή κειμένου, η μείωση του πεδίου εφαρμογή της γνωμοδότησης. Δεν θα συμφωνήσω με αυτές θα προτείνω να τις καταψηφίσουμε. Βάσει πάντως των τροπολογιών εκείνων που προσθέτουν στοιχεία Προσπάθησα και κατέληξα σε τρεις συμβιβαστικές τροπολογίες που θα συζητήσουμε την Τετάρτη για να τις καλύψω αυτές τις τροπολογίες. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί. Πάντως το μόνο θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τους Σκιώδης και να το πω ήδη εδώ, είναι ότι επίσημα πρόκειται για μια γνωμοδότηση στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων όσον αφορά την εφαρμογή της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πολλές τροπολογίες που υποβλήθηκαν έχουν να κάνουν περισσότερο με το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να φροντίσει να τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα στις χώρες μέλη. Υπήρχαν πολλοί ακραίοι. Να μην ξεχνάμε όμως ποιο είναι το αντικείμενό μας εδώ. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε για να προχωρήσουμε γρήγορα και να πετύχουμε συνένεση τελικά. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ, Ντένις. Τώρα, ποιος θέλει το λόγο. Κάποιοι έχουν ζητήσει να μιλήσουν, κάποιοι σκιώδεις. Σοσιαλιστές. Κριστίν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα αρχίσω ευχαριστώντας τους συναδέρφους που συνυπέγραψαν τις τροπολογίες μου. Δεν θα έρθω σε όλες, αλλά θα επιμείνω σε κάποια στοιχεία που για μα είναι πολύ σημαντικά. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά την εφαρμογή της χάρτας από τις χώρες μέλη. Γιατί το άρθρο 51 ακριβώς λέει ότι εφαρμόζεται στις χώρες μέλη. Οπότε πρέπει αυτό το άρθρο να διευκρινιστεί και η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής προς όφελος όλων των πολιτών. Και έχω μια τροπολογία για τις θετικές υποχρεώσεις που προβλέπει η χάρτα αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δρά άπαξ και τα δικαιώματα τα οποία γράφονται στη χάρτα απειλούνται. Υπάρχει μια σημαντική και ενδιαφέρουσα τροπολογία, αριθμό 38, για ένα μηχανισμό που μας επιτρέπει να παρακολουθούμε τι γίνεται με τα θεμελιώδη δικαιώματα στις χώρες μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Τέλος, έχω και μια τροπολογία για την απόφαση της Πολωνίας στη συνεδρίαση των Υπουργών δικαιοσύνη, όπου αντιτάθηκε στην πρόταση του Συμβουλίου για την εφαρμογή τη χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και διαβάζοντα τι 67 τροπολογίες βλέπω ότι είμαι η μόνη που αναφέρομαι σε αυτό. Καλό είναι όμω να ε, σημειώσουμε ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο δρούμε. Ένα δύσκολο πολιτικά πλαίσιο. Γενικά οι τροπολογίες ε, με ενθαρρύνουν αυτές που έχουν υποβληθεί και είναι πολλές και από τους πρασίνους αλλά και από τον εισηγητή και ευχαρίστω να συζητήσουμε στην ε, συνεδρίαση που οργανώνεται με τους υπόλοιπους σκιώδες για τις τροπολογίες αυτές. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ Κριστίν. ECR, Γιούρεκ. Παρακαλώ κύριε Γιούρεκ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρόεδρε, οι τροπολογίες που εμείς έχουμε υποβάλει επικεντρώνονται σε δύο τομείς κυρίως. Πρώτα απ' όλα, πρόκειται για την αρχή της επικουρικότητας. Πρέπει να επιμείνουμε, να ξέρουμε ποιες είναι οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κάτι γενικό, αλλά είναι και ειδικό σε αυτή την περίπτωση. Και ελπίζω να βρούμε τρόπο με συμβαστικές τροπολογίες, με συμβασμούς, να έχουμε μια καλή έκθεση προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πάντως. Ενώ και μιλάω για τη δικαιώματα των γονιών όσον αφορά τις επαφές τους με τα παιδιά τους. Ξέρουμε στη Γερμανία το Jungendamm, το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει εκεί, αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Υπάρχει και το άρθρο 24 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ελπίζω οι τροπολογίες που μιλούν για τα δικαιώματα των γονιών όσον αφορά τις σχέσεις τους με τα παιδιά τους και τις επαφές με τα παιδιά τους να βρουν σύμφωνο τους συναδέρφους και να εγκριθούν ώστε να συμπεριληφθεί και αυτό το θέμα ε, στην ε, τελική γνωμοδότηση. Ελπίζω να μπορέσουμε να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριο Τερικάμπρας, παρακαλώ, εκ μέρου των Πρασίνων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ. Χαίρομαι που βλέπω ότι ο συνάδελφο Ντεγιόγκα χαίρεται που βλέπει τους συναδέρφους που έχουν έρθει εδώ στην αίθουσα για την εκθεσή του. Σας ευχαριστώ που το εκτιμάτε. Εκτιμάτε την παρουσία μας εδώ. Πρόεδρε, Ευχαριστώ για το σχέδιο γνωμοδότησης του συντάκτη που καλύπτει πολλές από τις δικές μας ανησυχίες. Σήμερα είδαμε και τις συμβαστικές τροπολογίες που προτείνει ο εισηγητής. Και, από... και με μια πρώτη ματιά υπάρχει το θέμα της ίδιας της εφαρμογής της χάρτας θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το γεγονός ότι εφαρμόζεται μόνο σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον ε, βέβαια πρόκειται συγχρόνως για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου, θεωρούμε ότι δεν είναι αρκετό και δεν ικανοποιεί πολλούς ε, συμπολίτες μας, όπως εμάς για παράδειγμα. Γιατί μια τέτοια κατάσταση δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη αποξένωση των πολιτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα έπρεπε να σκεφτούν να ενισχυθεί περισσότερο και να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της χάρτας αυτής. Είμαι βέβαιος ότι από κοινού με τους σκιώδει θα καταλήξουμε σε μια πάρα πολύ καλή γνωμοδότηση. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τερικάμπρα. Υπάρχει κάποιο άλλο όχι. Ωραία. Ευχαριστώ Ντανής. Εγώ την παρακολουθούσα την νομοδότηση, ήμουν εδώ. Ε, είναι ενδιαφέρον ότι κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι τεχνικό, μια γνωμοδότηση στην ΑΦΚΟ, έχει 67 τροπολογίες. Είναι ενδεικτικό αυτό. Όλα είναι ενδιαφέροντα πια στην Επιτροπή μας. Ε, είναι αφέλεια να σκεφτόμαστε ότι θα υπάρξει κάτι χωρίς τροπολογίες. Όπως είπε και η Κριστίν. Και έγινε λοιπόν πολύ ενδιαφέρουσα η γνωμοδότηση. Έχουμε την ψηφοφορία που είναι προγραμματισμένη για τον Ιανουάριο. Θέλετε να πείτε κάτι. Όχι, να πω μόνο ότι η Κριστίν είχε δίκιο όταν είπε ότι οι συνεδρίες των σκιωδών είναι αύριο και όχι την Τετάρτη. δεν είναι πρόβλημα. Εγώ την αναμένω. Ωραία, σας ευχαριστώ. Ε, μεγάλη αίθουσα. Γι' αυτό μοιάζει άδεια. Καταλαβαίνετε. Στο άλλο κτίριο κάνουμε μπουγιο. Μην να κάνετε έτσι. Σημείο 5. Εφαρμογή των διατάξεων της συνθήκης που αφορούν την ενισχυμένη συνεργασία. Λοιπόν, έχουμε συναδέλφους από την Επιτροπή ΑΦΚΟ. για να αξιολογήσουμε τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε από τη χρήση αυτού του νέου μηχανισμού. Η Επιτροπή μας θα γνωμοδοτήσει μια που είναι αποκλειστική της αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η δημιουργία της οποίας βασίζεται στο άρθρο 86 της συνθήκης. Χαίρομαι λοιπόν που ήρθε ο εισηγητής, ο κύριος Σντεχόφσκι. Έχετε τον λόγο αγαπητέ. Χαίρομαι ιδιαιτέρως και εγώ που είναι ο πρόεδρος εδώ. Θα παρουσιάσω την έκθεση μου λοιπόν γρήγορα. Τώρα θα μιλήσω την τσεχική. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους ε, που μου έστειλαν τις πρώτες τους παρατηρήσεις την τελευταία εβδομάδα την ε, Τρίτη επεξεργαστήκαμε το κείμενο και το στείλαμε σε όλους τους συναδέλφους. Βασικό στόχος είναι να γίνει το σύστημα ελκυστικό για όλα τα κράτη-μέλη. Και βεβαίως ακριβώς είδαμε το πως ε, μπορούμε να κινηθούμε γρηγορότερα στα κράτη-μέλη. Το πλαίσιο ενισχυμένης ε, συνεργασίας δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί και ακριβώ προσπαθούμε να δώσουμε όλα αυτά τα κίνητρα έτσι ώστε η υπηρεσία αυτή να ενισχυθεί όπως και να ενισχυθεί και να η συνεργασία απευθύνω έκκληση στα κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν ενταχθεί ακόμα να το κάνουν μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου λοιπόν μία η ώρα θα πρέπει να υποβληθούν ε, οι τροπολογίες σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας σας ευχαριστώ αγαπητέ Κοιτάω να δω αν θέλει κάποιος τον λόγο. Όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, η προθεσμία είναι σε 7 Δεκεμβρίου, μία η ώρα το μεσημέρι. Ευχαριστώ. Προχωράμε πάρα πολύ γρήγορα, συναδελφοί, και περνάμε στο σημείο 6. Α, εγώ είμαι ο εισηγητής, μάλιστα. Να το προχωρήσουμε. Οπότε... Συνάλληφοι, θα προχωρήσουμε στη μέση διαταξία, γιατί έχουμε πολλές ψηφοφορίες. Είμαστε λίγο μπροστά από το πρόγραμμα. Ξέρω πως οι συνάδελφοι έρχονται την ώρα που είναι το θέμα που τους ενδιαφέρει και μετά αν προχωράμε γρήγορα το χάνουμε, αλλά τι να κάνω τώρα. Σας πειράζει να κάνουμε ένα διάλειμμα λίγων λεπτών. I'm just going a, I'm just going a bit too fast. Um... Γιατί είπε, πήγαμε πάρα πολύ γρήγορα. Και κάποιοι συνάδελφοι έρχονται. Ε, είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει μαζική προσέλευση στο επόμενο θέμα. Σας ευχαριστώ. We'll, we'll resume in about five, five minutes if you don't mind. Um, Αγαπητοί συνάδελφε, χαίρομαι που επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Η Δευτέρα είναι και δύσκολη ημέρα. Ο κόσμος ε, έρχεται με το αεροπλάνο και είναι δύσκολο αυτό. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα με το σημείο 6. Ένα ψήφισμα αφορά μια παρουσίαση της Κομισιόν. Όχι, δεν είναι παρουσίαση. Το θέμα, εν πάση περιπτώσει, είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα ανθρώπων αφρικανικής καταγωγής και όπως ξέρουμε ε, είναι αυτό. Αρμοδιότητα της Επιτροπής μας. Έχουμε αρμοδιότητα για τα θέματα αυτά που αφορούν την καταπολέμηση κάθε είδους ε, διάκρισης ε, πλην των σεξουαλικών και των εργασιακών. Έχουμε αφιερώσει όμως ε, συγκεκριμένα χρόνο και ειδική προσοχή στην κατάσταση ανθρώπων αφρικανικής ε, καταγωγής και ειδικά το θέμα του ρατσισμού και της διακριτικής μεταχείρισης. Και θα ήθελα τώρα να ευχαριστήσω την συνάδελφο την κυρία Κιέγγε που μας ενέπνευσε για αυτό παρά το ότι γίνεται προς το τέλος της εντολής είναι κάτι το πολύ επίκαιρο και άργησε κιόλα και χαίρομαι που επιτέλους το κάνουμε το σχέδιο ψηφίσματος αναφέρεται σε μελέτες όπως αυτές που δημοσίευσε η Ένωση Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αλλά και η σχετική υπηρεσία την προηγούμενη εβδομάδα που αναφέρει σαφώς ε, το φαινόμενο μιλάει για ζητήματα ρατσισμού και διακρίσεων και ζητάει να καταπολεμηθούν και επίσης ζητάει επίσημη αναγνώριση της ιστορίας ε, των Αφρικανών στην Ευρώπη και να δούμε την κοινή μας ιστορία και να ενθαρρυνθεί η πολιτική συμμετοχή των ανθρώπων αφρικανικής ε, καταγωγής. Ε, μια απλή ματιά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Νομίζω αυτό αποδεικνύει ότι χρειάζεται αυτό. Ειδικά όσον αφορά την πολιτική τους εκπροσώπηση αλλά και γενική εκπροσώπηση στα θεσμικά όργανα αυτό ισχύει γενικώ για τους εγχρώμους, αλλά ειδικώ όσον αφορά τους ανθρώπους αφρικανικής καταγωγής. Αυτά τα αναφέρει το σχέδιο ψηφίσματος, ε, Όπω επίση και τα άλλα ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ναι, και ε, για τους ανθρώπους αυτούς ε, το σχέδιο αυτό εγκρίθηκε από τους συντονιστές ε, και θα ολοκληρωθεί η συζήτηση με μια προφορική ερώτηση που επίσης εγκρίθηκε από τους συντονιστές ε, και την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ την προηγούμενη εβδομάδα. Θα υποβληθούν αυτά στην διάσκεψη των Πρόεδρων ε, για να περιληφθούν στην Ολομέλεια του Ιανουαρίου με συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 128. Χαίρομαι λοιπόν που είναι στην ημερήσια διάταξη και αναγνωρίζουμε αυτήν την μόρφη διακριτικής μεταχείρισης σε αυτή την δύσκολη καμπή. Μετά από αυτά, ήθελα να ρωτήσω τους και ηγητές αν έχουν κάτι να πούν και μετά αν έχουμε κάποιον άλλον που θα ήθελε να σχολιάσει. Δεν είναι εδώ η συντονίστρια του ΕΛΚ. Οπότε θα ζητήσω από την ε, ε, εισηγήτρια των Σοσιαλδημοκρατών, την Σεσίλ, να μας πει δύο λόγια. Έχετε τον λόγο. Σε ευχαριστώ, Κλόντ. Και θα ήθελα ειλικρινά να ευχαριστήσω εσένα καταρχάς γιατί είσαι πρόεδρος της Επιτροπής αυτής και ασχολήθηκες με την όλη διαδικασία που οδήγησε σε αυτή την πρόταση ψηφίσματος. Όχι μόνο στα πλαίσια της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, αλλά και για όλες τις προσπάθειες που καταβάλεις καθημερινά στην όλη αυτή διαδικασία προκειμένου να καταλήξουμε σε μία Ευρώπη η οποία θα σέβεται τα δικαιώματα όλων. ευχαριστήσω βέβαια και όλους που συμμετείχαν από όλες τις πολιτικές ομάδες όλους αυτούς οι οποίοι πραγματικά συνέβαλαν στο να αναγνωριστούν τα δικαιώματα αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή μια επονίδιστη κατάσταση όσον αφορά την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα φαινόμενα ρατσισμού, ξενοφοβίας, φαινόμενα τα οποία παίρνουν πολλές διαφορετικές μορφές. Δεν είναι μόνο φαινόμενα μίσους και ρατσισμού κατά των ανθρώπων αφρικανική καταγωγή, αλλά έχουμε διακριτική μεταχείριση και μίσος που παίρνουν και πιο έμεσες μορφές. Ουσιαστικά αναφερόμαστε εδώ πέρα σε ένα είδος διαρθρωτικού ρατσισμού που βάλει κατά των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είδαμε και τις επιθέσεις οι οποίες έλαβαν χώρα κατά των ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή και εν γέννη κατά όσων είναι μαύρων. Νομίζω λοιπόν, στη Ματσαράτα για παράδειγμα της Ιταλίας είχαμε τέτοια φαινόμενα όπου ο Λούκα Τράινι στα, στα, στο μέσο, στα μέσα του δρόμου, σε έναν δρόμο, στη διάρκεια μιας διαδήλωσης, είπε ότι θα ήθελα να σκοτώσω ως το δυνατόν περισσότερους μαύρους. Νομίζω λοιπόν ότι μετά από τέτοια φαινόμενα, μετά από τέτοια επεισόδια, θα πρέπει πραγματικά να παρακολουθήσουμε και όλα αυτά τα οποία ακολούθησαν. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια έκθεση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, όπου ξεκάθαρα οριοθετεί το πλαίσιο εκείνο το ευρωπαϊκό για την καταπολέμηση τη παραβίαση των ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών με αφρικανική καταγωγή. Με την έκθεση αυτή δεν έχουμε μόνο μια καταγγελία των κακών κειμένων, αλλά έχουμε επίση και συγκεκριμένε συστάσει για το πώ θα αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό, συγκεκριμένε κατευθύνε γραμμέ, οι οποίε θα πρέπει να ακολουθήσουμε στο μέλλον. Εγώ πήγα σε ορισμένα κράτη-μέλη, για παράδειγμα στην Γαλλία και στην Αγγλία, όπου είδα ότι υπάρχει εκεί πέρα μια πλήρη συνειδητοποίηση από πολλέ κοινότητε πολιτών προκειμένου να υπάρχει μια καλύτερη συμμετοχή κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και πολιτική των ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι αλλάζει η όψη της Ευρώπης πλέον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι άνθρωποι με αφρικανική καταγωγή να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες κοινωνίας μας και να μπορούν να εκπροσωπηθούν και να εκφραστούν ελεύθερα. Νομίζω λοιπόν ότι η πρόταση αυτή ψηφίσματος μπορεί να οδηγήσει μια πιο πολυπολιτισμική ισότιμη, δίκαιη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Μια κοινωνία που δεν θα υπάρχει κανένα χώρος για αυτό το ρατσιστικό μίσος. Νομίζω ότι τέτοια εργαλεία, τέτοια μέσα όπως το ψήφισμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικά προκειμένου να καταφέρουμε να δυναμώσουμε μια κοινωνία η οποία θα πρέπει να είναι πολυπολιτισμική. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Εν γέννη πρέπει να πούμε ότι το ζήτημα του, της διακριτικής μεταχείρισης κατά των ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή, με καταγωγή επίσης από την, γενικότερα την Αφρική, την Καραϊβική, θα πρέπει να εξεταστεί και στην αγορά εργασίας αλλά και στην πρόσβαση στη στέγαση καθώς επίσης και σε άλλες υπηρεσίες. Αναφέρονται όλα αυτά στην πρόταση ψηφίσματος και είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη και τα φαινόμενα αυτά, τα κρούσματα ρατσισμού τα οποία έθιξες και εσύ Σεσίλια στην Ιταλία. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει η κυρία Γερόκα. Να σα συγχαρώ και εγώ για την εκθεσή σα, αυτή κύριε Πρόεδρε και να ευχαριστήσω επίση και την κυρία Κέγγε η οποία έχει αναλάβει πολύ δραστηριό ρόλο και βρέθηκε πραγματικά στην πρώτη γραμμή όσον αφορά τα ζητήματα αυτά, ιδίω για του ανθρώπου με αφρικανική καταγωγή. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να ενισχύσουμε, να δυναμώσουμε του ανθρώπου αυτού, οι οποίοι ζουν στην Ευρώπη και οι οποίοι θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στις κοινωνίες μας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ιδιαίτερα καταρτισμένοι, είναι ε, άνθρωποι οι οποίοι έχουν τόσο την ε, γνώση και την πείρα που έρχεται από την ε, χώρα από την οποία κατάγονται, αλλά έχουν ζήσει και στην Ευρώπη πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι μπορούν να γεφυρώσουν πραγματικά πάρα πολύ του δύο αυτού κόσμου. Πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να ενισχύσουμε του ανθρώπου με αφρικανική καταγωγή που ζουν στην Ευρώπη. Παράλληλα όμω, είναι πολύ σημαντικό, όπω είπατε κι εσεί, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταφέρει να αποτελέσει υπόδειγμα, να προωθήσει βέλτιστες πρακτικές, να εμπλέξει περισσότερους εμπειρογνώμονες, καθώς επίσης και περισσότερους ανθρώπους με αφρικανική καταγωγή που ζουν στην Ευρώπη. Λυπάμαι όταν βλέπω ότι υπάρχουν ε, χώρες όπως αυτές της Βόρειας και της Ανατολικής Ευρώπης που δεν στέλνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ευρωβουλευτές με αφρικανική καταγωγή. Επίσης, ο, ρόλο, ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικός. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε ότι ε, όλοι οι άνθρωποι με αφρικανική καταγωγή, ιδίω οι πιο ευάλωτοι, οι πιο φτωχοί, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα απαραίτητα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Νομίζω όμως ότι ανάλογη κατάρτιση θα πρέπει να έχουμε και για τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης που θα πρέπει να προβάλλουν μια πιο θετική εικόνα των ανθρώπων αυτών. Επίσης, πρέπει να ενισχύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα και την προστασία των δικαιωμάτων αυτών για τους ανθρώπους με αφρικανική καταγωγή. Σαφώς χρειαζόμαστε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμα και καλύτερη εκπροσώπηση των ανθρώπων αυτών προκειμένου να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο να ζουν καλύτερα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να υπάρχει καλύτερη αντιμετώπιση των χωρών καταγωγής τους. Αν δεν τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη, δεν νομίζω ότι μπορούμε επικοδομητικά να συζητήσουμε ζητήματα που άπτονται της μετανάστευσης. Όπως ε, λέει και η έκθεση αυτή, θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στις μελλοντικέ λύσεις για αυτούς που έχουν αφρικανική καταγωγή και ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Σας ευχαριστώ. Και εμεί σα ευχαριστούμε πολύ, Ολίβια. Και οι υπόλοιποι σκιώδει ηγητέ, όπω η Άννα Μαρία Κοράτσα Μπίλτ, ο Λί Μισελ, η Μαλίν Μπιόρκα από την ΚΟΕ, μου έχουν πει ότι ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την πρόταση αυτή ψηφίσματο. Κατά πάση πιθανότητα θα πρέπει να ταξιδεύουν και Δευτέρα απόγευμα, μια δύσκολη μέρα. Πάντως ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το περιεχόμενο τη πρώτης αυτή ψηφίσματο. Μπίργκιτ, θέλετε τον λόγο. Θα έλεγα τώρα τους άλλους ότι αν δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο θα το κλείναμε, αλλά προφανώς έχετε το λόγο. ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, μια σύντομη παρατήρηση έχω να κάνω. Πράγματι, συνάδελφος έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα και πρέπει ακριβώς να αλλάξουμε οπτική γωνία ε, δεν θεωρώ δηλαδή ότι όλοι οι άνθρωποι αφρικανικής ε, καταγωγής ε, που ζουν εδώ πέρα χρειάζονται βοήθεια και στήριξη. Τουλάχιστον όχι στον βαθμό που χρειάζονται κάποιοι άλλοι. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να σταματήσουν οι διακρίσεις να τους δεχτούμε ως ανθρώπους ε, και να τους μεταχειριστούμε ανάλογα και όχι χειρότερα λόγω καταγωγής. Το ίδιο ισχύει και για το θέμα των εξελίξεων στις χώρες σε προέλευση. Βεβαίω είναι πάντα ευπρόσδεκτη η βοήθεια, αλλά πολλές εξελίξεις στις αφρικανικές χώρες θα ήταν πολύ καλύτερες εάν κάναμε πολιτική με την Αφρική όχι πάντα αποκλειστικά υπό τη σκοπιά του τι είναι καλό για εμάς, αλλά να δώσουμε την ευκαιρία σε αυτούς τους ανθρώπους να αναπτύξουν δική τους βιομηχανία, οικονομία και πολλαπλασιασμό της αξίας. αντί να αγοράζουμε φτηνές πρώτες και να πουλάμε ακριβά προϊόντα. Πρέπει ακριβώς να δούμε και την σκοπιά που έχουμε για την Αφρικανική Ήπειρο. Αλλιώ δεν θα επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ. Αυτό το οποίο θα τόνιζα εγώ το ψήφισμα αυτό είναι ότι δεν αφορά την Αφρική. Α, μιλάμε για Αφρικανούς που είναι εδώ, και αιώνες και εργάζονται και δουλεύουν μεταξύ μόνο και θέλουν απλά να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού και αντιλαμβάνονται ότι έχουμε μία κορύφωση της, α, των διακρίσεων α, και πριν από 20 χρόνια που ήρθα εγώ υπήρχαν περισσότεροι Αφρικανοί ευρωβουλευτές τα πράγματα δηλαδή χειροτερεύουν και αυτό φαίνεται και σε κάποιες αγορές εργασίας και σε κάποια άλλα ζητήματα αστυνομία δικαστηρίων που θα έπρεπε να βελτιώνεται η κατάσταση. Και ανέφερε η Κυριακή Έγκαι ζητήματα όσον αφορά την άνοδο του λαϊκισμού. Χαίρομαι λοιπόν που φέραμε αυτό το ψήφισμα και όταν ξεκινήσαμε αναρωτιόμουν αν θα μπορούσαμε να κάτι και, και ευχαριστώ τη γραμματεία που μας έδωσε αυτή την δυνατότητα Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι και κυρίως την Σεσίλ Κιέγγελ που μας ενέπνευσε με την δουλειά της και βεβαίω χάρη ε, στη δουλειά της υπηρεσίας θεμελιωδών δικαιωμάτων σας είπα το χρονοδιάγραμμα θα εγκριθεί το σχέδιο ψηφίσματος στις 10 Δεκεμβρίου και θα το συζητήσουμε και θα το ψηφίσουμε στην Ολομέλεια, στην πρώτη Ολομέλεια του Ιανουαρίου. Ελπίζω να είναι εκεί κάπως πιο έντονη η συζήτηση από ό,τι τώρα. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Ευχαριστώ όσους συμμετείχαν. Περνάμε στο σημείο 7. Ακριβώς την ώρα εκθεσία από την αναφορά από την αποστολή μας για το κράτος δικαίου στην Πολωνία 19 με 21 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, να αναφέρω τις τεχνικές πτυχές. Πριν περάσω στις λεπτομέρειες. Λοιπόν, συνάδελφοι, η αποστολή αυτή στην ε, Βαρσοβία θα σας πω τα ονόματα των συναδέλφων γιατί ήταν μια ευαίσθητη αποστολή είχε τεχνικές πτυχές επικεφαλής ήμουν εγώ η κυρία Σαρτζεντίνη από τους Πράσινους είχαμε τον κύριο Τόμασεύσκι τον κύριο Έγγελ τον κύριο Μπέι την κυρία Σπινέλη και την κυρία Μπερζερόν. Έχει οριστικοποιηθεί το σχέδιο έκθεσης ε, σε συνεργασία με τα μέλη της Αποστολής και επιπλέον ήρθαμε σε επαφή με τους συνομιλητές μας ε, στη Βαρσοβία και έχουν σχολιάσει. Κάποιοι μάλλον έχουν σχολιάσει, κάποιοι δεν έκαναν κάποια σχόλια. Τέλος, οι πολωνικές αρχές είχαν μία εβδομάδα καιρό για να σχολιάσουν ε, το σχέδιο έκθεσης, πρέπει να το αναφέρω αυτό. Την Τετάρτη έλαβα μια επιστολή από τον Πολωνό πρέσβη με κάποια ειδικά και γενικά σχόλια. Και θα επισυναθεί η επιστολή αυτή όπως και η αποστολή μου. Και η ε, απάντησή μου, με συγχωρείτε. Τώρα, να σας πω ποιοι ήταν οι στόχοι, ποιες συναντήσεις είχαμε και τα βασικά ευρήματα. στόχος της αποστολής ήταν να αντιληφθούμε καλύτερα τις μεταρρυθμίσεις της δικαιοσύνης που κάνουν οι πολωνικές αρχές οι στόχοι της κατάστασης αυτής και ο αντίκτυπος στο κράτος δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 7. Συναντηθήκαμε με μέλη της Βουλής, της Γερουσίας, πολιτικά κόμματα, εκπροσώπους ε, του ΟΑΣΕ, νομικούς, δημοσιογράφους και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε λοιπόν όλους τους συνομιλητές, ε, κάποιους από τους οποίους συναντήσαμε ξανά την προηγούμενη εβδομάδα, με ευκαιρία της ακρόασης, για το ότι ήταν διαθέσιμοι. Κατέβαλε η αντιπροσωπεία κάθε προσπάθεια για να συναντηθεί με όσο δυνατόν περισσότερους συνομιλητές λυπούμεθα για το ότι κάποιες συναντήσεις δεν έγιναν και παρουσιάζουμε ποιες ήταν αυτές ως επικεφαλής εγώ ζήτησα να συνδεθώ με τον πρόεδρο, τον πρωθυπουργό τον υπουργό δικαιοσύνης και τον αρχηγό του κόμματος ε, δικαίου και δικαιοσύνης Κανένα συνάντησα κανέναν από αυτούς. Έλαβα μία απάντηση από τον Πρωθυπουργό στις 19 Δεκεμβρίου που μας είπε ότι κολλείεται. Όπως είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας αντιλαμβάνουμε ότι είναι απολύτως ε, θεμητό οι πολωνικές αρχές να μεταρρυθμίσουν την δικαιοσύνη και άκουσα πολύ προσεκτικά τις εξηγήσει που έδωσαν οι αρχές. Όμως θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι μετά από την ιστορική ένταξη της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Πολωνοί δικαστές δρούν ως Ευρωπαίοι δικαστές και έχουν καθήκον να διασφαλίσουν μια δίκαιη και αμερόληπτη εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Έχοντας λοιπόν ακούσει όλους τους συνομιλητές μας, παρουσιάσαμε τα κυριότερα ευρήματα με τα οποία συμφώνησαν όλα τα μέλη εκτός από τον κύριο Τόμασεύσκη του ΙΣΙΑΡ, και τον κύριο Μπέι του ΙΕΝΕΦ. Οπότε η αντιπροσωπεία ανησυχεί για το σωρευτικό αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης ε, που γίνεται τα τελευταία τρία χρόνια και επηρεάζει το Συνταγματικό Δικαστήριο, τα Τακτικά Δικαστήρια, το Εθνικό Συμβούλιο Δικαιοσύνης, το Ανώτατο Δικαστήριο, τα οποία μαζί φαίνεται ότι αποτελούν ένα σοβαρό κίνδυνο για το κράτος δικαίου στην Πολωνία. Επιπλέον η αντιπροσωπεία ανησυχεί μεταξύ άλλων για την σύνθεση και λειτουργία του Συνταγματικού Δικαστηρίου, τη δημοσίευση ορισμένων αποφάσεών του, την μεταρρύθμιση των νέων δικαστηρίων και τις ε, συνεχείς ε, και συστηματικές επιθέσεις σε δικαστές ε, με πειθαρχικές διαδικασίες, ειδικά κατά των δικαστών που είναι κατά των μεταρρυθμίσεων και την παραπομπή και όσων παραπέμπουν προδικαστικά ερωτήματα στο ΔΕΚ και τις μεταθέσεις αυτών. Η συσσόρευση των εξουσιών επίσης στο επίπεδο του Υπουργού Δικαιοσύνης, ε, κάτι το οποίο πριν δεν υπήρχε. Ένα άλλο θέμα είναι η σύνθεση και οι αρμοδιότητες του νέου Συμβουλίου Δικαιοσύνης, ε, το οποίο αφορά το καστός εκλογών, το καστός συνταξιοδότησης ε, των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου, που σήμαινε ότι διακόπηκε η θητεία του Προέδρου παρά το το Σύνταγμα προβλέπει εξαετή θητεία και αφορά αυτό 27 από τους 72 δικαστές που αποτελούν αυτή τη στιγμή το Συνταγματικό Δικαστήριο. Ένα άλλο θέμα ήταν η διακριτική ευχέρεια του Προέδρου και του Υπουργού Δικαιοσύνης να παρατείνουν την θητεία δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και των Τακτικών Δικαστηρίων χωρίς να το αιτιολογήσουν ούτε δυνατότητα των δικαστών έχουν κάποια αντίρρηση μετά. Υπήρχε νομική αβεβαιότητα και η διαδικασία εφέσεων ε, Επίσης υπάρχει νομική αβεβαιότητα που αφορά τις ε, μελλοντικέ εκλογές ε, για την έλλειψη ανεξαρτησίας ή έλλειψη δημόσιας διαβούλευσης κατά τη διάρκεια των νομοθετικών διαδικασιών, ε, οι επιδεινόμενες συνθήκες λειτουργίας των ΜΜΕ, παραδείγματο χάρη πρόσβαση σε πηγές ε, της ε, κυβέρνησης, παρά το ότι υπάρχει μια σχετική ελευθερία των ΜΜΕ, υπάρχει ένα πολλωμένο τοπίο στα ΜΜΕ, Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένες συνθήκες που επιδεινώνονται. Οι συνθήκες επίσης λειτουργίας των ΜΚΙΟ, μειωμένη χρηματοδότηση, ε, αυξημένα διοικητικά βάρη, παρά το ότι ανθεί η κοινωνία των πολιτών. Ζητήματα για τις γυναίκες, ε, ε, ειδικά στις περιφέρειες για βασικά αναπαραγωγικά δικαιώματα, έλλειψη πρόσβαση πληροφορία, το χάπι τη επόμενη μέρας, προγεννητική έλεγχη κτλ. Έλλειψη εφαρμογής, ή συστάσει τη Επιτροπής της Βενετίας για το πλαίσιο κατσουκαίου. Και βεβαίως έχουμε το μέλος του ECR τον κύριο Τομασεύσκη που εξαιρείται από τα συμπεράσματά μας ε, και με την αξία του κύριου Τομασεύσκη έχουμε την ανησυχία της Επιτροπής για το ότι παραβιάζονται κάποιες βασικές αρχές του κοινού μεταξύ των οποίων η ανεξαρτησία της δικαιοσύνη, η δίκαιη δίκη και άρα συμφωνούμε με την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θεωρεί ότι υπάρχει σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης του κρατζουκαίου από τις αρχές της Πολωνίας. Αυτή είναι η εκθεσή μου. Όπως σας είπα θα επισυναυθεί και η επιστολή του Πολωνού πρέσβη και θα ήθελα τώρα να ζητήσω από τους συναδέλφους να σχολιάσουν. Η κυρία Σαρτζεντίνη ήταν επίση ε, στην αντιπροσωπεία και θα ήθελα να σχολιάσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συμμετείχα και εγώ στην αντιπροσωπεία αυτή και χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν μετά τη βδομάδα μετά την ψηφοφορία που είχαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την έκθεση για την Ουγγαρία. Και αυτό που βρίσκω ότι είναι πολύ σημαντικό είναι ότι δημιουργήσαμε μια τάση για να κάνει όσον αφορά το άρθρο 7 τη δουλειά σου στα σοβαρά, πά στη χώρα, συναντάς τους αξιωματούχους, τον κόσμο, ε, στα διάφορα θεσμικά όργανα, στην κοινωνία των πολιτών, δικηγόρους κλπ. Επίσης να σας πω ότι μία μέρα το πρωί είχαμε επίσκεψη σε ένα νομικό όργανο το οποίο προεδρεύει την πρόσληψη και την απόλυση δικαστών. Και υπάρχουν και βουλευτές εκεί. Και το απόγευμα μιλήσαμε με τη Γερουσία και κάποιος γερουσιαστής μας είπε «Χαιρόμαστε που σας ξαναβλέπουμε γιατί και σήμερα το πρωί ήμασταν μαζί σας στην πρωινή σας επίσκεψη σε αυτό το ε, Συμβούλιο για τον έλεγχο των δικαστών». Αυτό ακριβώς είναι απόδειξη του προβλήματος που έχουμε να αντιμετωπίσουμε εκεί. Ένα άλλο σχόλιο τώρα, όχι τόσο για τα συμπεράσματα, γιατί συμφωνώ με τα συμπεράσματα. Αυτό που εκτίμησα ιδιαίτερα είναι ότι εξετάσαμε πολλά και διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, θεμελιώδη δικαιώματα κτλ. Και δεν περιοριστήκαμε στενά ε, στο άρθρο 7. Συναντηθήκαμε με δημοσιογράφους, για παράδειγμα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι δεν μπορείς να απλοποιήσεις τη διαδικασία του άρθρου 7 σε ένα στενά δικαστικό θέμα και να αναθέτεις, να βάζεις ευθύνε στους ώμους κάποιου άλλου, το καλό νέο είναι ότι η πολωνική κυβέρνηση αποφάσισε να αλλάξει την νομοθεσία τη όσον αφορά την ηλικία συνταξιοδότηση στον Νότο Δικαστήριο των Δικαστών. Αλλά φοβούμε ότι και πάλι αυτό είναι ένα επιχείρημα για το Συμβούλιο που τα τρία τέταρτα της χρονιάς τους λέει να ένα άλλο θεσμικό όργανο να λαμβάνει την πρωτοβουλία, οπότε εμείς δεν έχουμε την ευθύνη. Εγώ Πιστεύω ότι αυτό θα ήταν ένα λογικό συμπέρασμα από πλευρά του Συμβουλίου. Έτσι καλλιώς η Επιτροπή είναι θεματοφύλακα των συνθήκων και μπορεί να φροντίσει, να προσφύγει κατά μιας χώρας έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι τηρείται το κεκτημένο. Οπότε, εκτίμησε ιδιαίτερα τη δυνατότητα που είχαμε ανταλλαγή απόψεων με όλους στην Πολωνία. Πολύ θετικό. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημιουργεί έτσι μία τάση στον τρόπο λειτουργίας της και άπαξ και προκύψει ξανά τέτοιο θέμα με κάποια άλλη χώρα, θα δείξουμε ότι να, αυτό το δρόμο ακολουθούμε, αυτή είναι η ρουτίνα μας και θα Πάμε να εξετάσουμε και εκεί ό,τι πρέπει να εξετάσουμε. Πρόεδρος, ωραία, άλλος κανείς θέλει το λόγο. Τίποτα προσωπικό για την Πολωνία, έτσι. Με τίποτα. Γιατί χάσαμε ένα Πολωνό στο μεταξύ. Λοιπόν, ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζούντιθ. Είναι ένα πολύ λεπτό και ενδιαφέρον θέμα και περίπλοκο βέβαια. Οπότε ευχαριστώ πολύ και τη γραμματεία της ΛΥΜΠΕ που βοήθησε για αυτή την επίσκεψη και όλες τις ομάδες βέβαια που συμμετείχαν. Η έκθεση συζητήθηκε στις πολιτικές ομάδες και εκτός από το ECR και το ΙΕΝΕΦ αν δεν υπάρχει αντίρρηση εγκρίνεται η έκθεση αυτή και θα προχωρήσει. Θα αποτελέσει δηλαδή την έκθεση της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πήγε στην Πολωνία. Παρακαλώ. Επιτρέψτε μου κάτι όσον αφορά τη διαδικασία. Θέλω να πω ότι πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό όλοι να ακούσουν για την έκθεση αυτή. Το άρθρο 7 τουλάχιστον οι διαδικασίες του άρθρου 7 πρέπει να ακολουθούνται πλήρως από όλες τις χώρες μέλη. Και κάθε φορά που εξετάζουμε την κατάσταση σε μια χώρα βάσει του άρθρου αυτού, οι επαφές να είναι με όλους και με την κοινωνία των πολιτών και με όλους. Αυτή τη φορά έγινε, αλλά να φροντίσουμε και στο μέλλον κάθε φορά που έχουμε κάτι τόσο σοβαρό να υπάρχει αυτή η επαφή με όλους. Αλλά το δεύτερο, ακριβώς επειδή υπάρχει άρθρο 7, θα πάει και πάλι στο Συμβούλιο, έτσι δεν είναι. Δηλαδή οι συγητές θα πάνε πάλι στο Συμβούλιο, έτσι. Το ίδιο έγινε και στην περίπτωση της Ουγγαρίας. Είναι πολύ σημαντικό. Κάποιος από τη ΛΥΜΠΕ, κάποιος συνάδελφος που παρακολουθεί το θέμα να πάει για να ακουστεί και αυτόν η φωνή. Η έκθεση θα συζητηθεί στο Συμβούλιο, ελπίζω, για να τα μάθουν και οι Υπουργοί και οι Πρωθυπουργοί και ο κύριος Σταγιάννη και ο Πρόεδρος να το ακούσει. Αλλά και εμείς, η Επιτροπή μας ΛΥΜΠΕ, να στείλουμε κάποιον για να δείξουμε ότι είμαστε επαγγελματίες, κάποιον που να μπορεί να εξηγήσει την κατάσταση. Ιδιαίτερα αν έχουμε μια, κάποιον από τη ΛΥΜΠΕ που να έρθει μαζί σας στο Συμβούλιο. Αυτό προτείνω. Έχοντας υπόψη μου τι έγινε στο Συμβούλιο με την Ουγγαρία, γι' αυτό το λέω. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Για το πρώτο, όσον αφορά τη συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Πάντα οι αντιπροσωπείες μας φροντίζουν να συναντηθούν με την κοινωνία των πολιτών και αυτή τη φορά η αντιπροσωπεία συναντήθηκε και με μη κυβερνητικέ οργανώσεις και ενημερώθηκαν και τους ζητήσαμε και σχόλια. Σχολίασαν, ε, έτσι τροποποίησαμε και εμείς την έκθεση γιατί τους τη στείλαμε για σχόλιά τους. Οπότε έχουμε υπόψη μας. Όσο και αν τεχνικά είναι κάπως δύσκολη η συμμετοχή όλων, παρόλα αυτά φροντίσαμε να ακουστεί και η δικιά του η φωνή στην έκθεσή μας. Τώρα για το διαδικαστικό που θέτεται, όντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινάει την διαδικασία κατά της Πολωνίας. Εμείς έχουμε τη σύμφωνη γνώμη, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για την Πολωνία. Γι' αυτό πήγε και την προσωπία, γι' αυτό έχουμε και αυτή την εκτενή έκθεση. Σας παρουσιάσαμε την έκθεση και θα συνεχίσουμε με αυτή τη διαδικασία. Ωραία. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς? Όχι από ό,τι βλέπω. Ωραία, άρα εγκρίνεται η έκθεση αυτή, αν δεν υπάρχουν ε, αντιρρήσει με την εξαίρεση των δύο ομάδων, όπως σας είπα. Τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι θα διακόψουμε μέχρι τις 4.30 για το επόμενο μας θέμα που είναι το σύστημα πληροφοριών Λίζα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και την υπομονή σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε. Λοιπόν, εξετάζουμε το σύστημα πληροφοριών. Ο κύριος Κοέλιο μας παρουσίασε ήδη στις 5 Νοεμβρίου το σχέδιο έκθεσής του με 483 τροπολογίες τελικά. Η προθεσμία ήταν 13 Νοεμβρίου. Έκτοτε, ο εισηγητή μου, του σκιώδε εισηγητέ δουλεύουν και συνεργάζονται προκειμένου να καταλήξουν σε συμβιβαστικέ τροπολογίε. Οπότε, θα δώσουμε το λόγο στον εισηγητή μα, τον κύριο Κοαγιό. Παρακαλώ κύριε Κοαγιό, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Σχεδόν 500 τροπολογίες έχουμε από όλες τις πολιτικές ομάδες μαζί. Τρεις συναντήσεις είχαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άλλες πέντε με τους σκιώδεις εισηγητές και πέντε ακόμα προβλέπονται μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Θα προσπαθήσω με τις σεβαστικές μου προτάσεις να καλύψω όσο γίνεται περισσότερες τροπολογίες. Κάποιες γραμμές είναι ξεκαθαρές ήδη. Οι περισσότερες πολιτικές ομάδες συμφωνούν με το σύστημα, να υπάρχει το σύστημα δηλαδή, με τα θέματα της διαλειτουργικότητας επίσης. Όσον αφορά την επιβολή του νόμου, συμφωνούν οι περισσότερες ομάδες με τον επιτρέπεται η πρόσβαση. Οι περισσότερες ομάδες επίσης συμφωνούν με το κείμενο που ήδη ισχύει. Οι περισσότερες ομάδες συμφωνούν και με το πλαίσιο προστασίας. Πρέπει να είμαστε όμως ξεκάθαροι. Πρόθεση ε, του σχεδίου αυτού είναι η προστασία ώστε να μπορούν να έχουν ελεύθερη διακίνηση όσοι έχουν θεωρήσεις μέσα στο σύστημα Σέγγεν. Οπότε είναι ένα φυσιολογικό βήμα τώρα το σύστημα φύσης. Είμαστε σε ένα στάδιο τώρα όπου συμφωνούν οι περισσότερες πολιτικές ομάδες και έτσι θα μπορέσουμε να αρχίσουμε διαπραγματεύσεις την επόμενη χρονιά υπό Ρουμανική Προεδρία. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε Κάρλος. Σκιώδες εισηγητές τώρα. Η Μαρή Κριστίν Βερζιά είναι η μόνη από τους κοιόδρους συζητητές που θέλει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πάντα χαίρομαι όταν συνεργάζομαι με τον κύριο Κοέγιο, ακόμα και όταν διαφωνούμε επί της ουσίας. Και φοβούμε ότι σε μένα οφείλονται πάρα πολλές τροπολογίες. Αλλά όπως το είπα και στη συνάντηση των σχεδόν, πολλές από τις τροπολογίες αυτές είναι τροπολογίες αρχής γιατί είμαστε κατά της επέκτασης ε, του συστήματος χωρίς όρια της χρήσης του συστήματος VIS. Με τις διάφορες έρευνες που έκανα, θυμήθηκα ότι αρχικά το VIS ήταν μόνο για τη Βόρεια Αφρική και μετά γεωγραφικά επεκτάθηκε στο σύνολο της Μέσης Ανατολής και των χωρών του κόλπου. Και τώρα μιλάμε για ολόκληρο τον κόσμο. Και γι' αυτό και εμείς είμαστε κατά αυτής της επέκτασης χωρίς όρια του συστήματος. Δημιουργούμε ένα ειδικό εργαλείο σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και σιγά σιγά το διαβρύνουμε. το επεκτείνουμε γεωγραφικά και όσον αφορά το περιεχόμενο των δεδομένων που χρησιμοποιούνται. Αυτό ακριβώς προτείνεται σήμερα. Όταν λοιπόν διαπιστώνω ότι το VIS έχει πάνω από 55 εκατομμύρια αιτήσει τη χρονιά που μας πέρασε και 40 εκατομμύρια δακτυλικά αποτυπώματα, σε τι κόσμο ζούμε με τόσα θέματα τα οποία διακυδεύονται. Μα δημιουργούμε εργαλεία τα οποία κινδυνεύουμε να τα δούμε να στρέφονται κατά των δημοκρατών και των προοδευτικών. Τελικά θα φακελώνουμε ακόμα και τα παιδιά. Για μένα, ένα παιδί είναι ένα παιδί, ο ανήλικο είναι ανήλικο μέχρι τα 18 του. Κάτω των 18 πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν μπορεί να χρησιμοποιούμε διάφορες ε, διατάξεις που να μπερδεύουν τα νούμερα, αν θα είναι από τα 12, από τα 16, από τα 13. Θα ήθελα λοιπόν διευκρινήσεις πάνω σε αυτά έτσι ώστε οι ανήλικοι, για παράδειγμα, να μην αποτελούν στόχο τέτοιων διαδικασιών. Επίσης, επαναλαμβάνω ότι είμαι κατά στην ε, βοήθεια από εξωτερικούς. Θα ήθελα αυτό να γίνεται με μέτρο και να υπάρχει ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο. Ξέρουμε ότι στις χώρες του Νότου, τις Αφρικανικές χώρες για παράδειγμα, οι πάροχοι υπηρεσιών αυτοί, οι εξωτερικοί, συμπεριφέρονται, θα έλεγα με τρόπο μάλλον καταστροφικό τελικά. Όσο πιο φτωχοί είμαστε, τόσο πιο ακριβά μας στοιχίζει η βίζα. Υπάρχει διαφθορά με δύο λόγια, δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ο ετών να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει την αίτησή του σε μη διπλωματική υπηρεσία. Επίσης, είμαστε κατά στην επέκταση των δεδομένων που συλλέγονται και των βιομετρικών δεδομένων κυρίως. Το σύστημα VIS πρέπει να παραμείνει ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για να εκδίδονται θεωρήσεις VIS και για τίποτα άλλο. Τότε πώς είναι δυνατόν να πολλαπλασιάζουμε τα δεδομένα τα οποία θα μπαίνουν σε αυτό το σύστημα από πολλέ και διαφορετικές αρχές, ακόμα και από κατασταλτικές αρχές. Συνεπώ, μένει πολλή δουλειά ακόμα για να πλαισιώσουμε το σύστημα αυτό με τρόπο ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί κακόβουλα ή σε ένα πλαίσιο που μπορεί στο μέλλον να αναπτυχθεί αρνητικά. Καλό θα ήταν να είμαστε σόφρονες και να χρησιμοποιούμε διάφορες ρήτρε ασφάλειας. Αλλιώ θα είμαστε σαν το βιβλίο του Όρουελ το 1984. Μην ξεχνάμε να κοιτάμε τι είναι αυτό που δημιουργούμε και που μπορεί να μας οδηγήσει. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε Μαρή Κριστίν. Άλλος κανείς θέλει το λόγο παρακαλώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ναι, πολύ σύντομα από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμεί προσβλέπουμε στην αρχή των διαπραγματεύσεων στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου. Ευχαριστούμε και τον εισηγητή και τους άλλους ευρωβουλευτέ. Είναι πολύ σημαντική πρόταση αυτή για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζουμε ακόμα σε αυτή τη θητεία να καταλήξουμε, να έχουμε μια συμφωνία. Οπότε περιμένουμε με ανυπομονησία την αρχή των διαπραγματεύσεων. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κάρλος, για να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα, τα σχόλιά σου. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, απλώς θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδες εισηγητές για τη βοήθειά τους. Έχουμε ένα πολύ επικοδομητικό κλίμα μεταξύ μας, μια πολύ καλή ατμόσφαιρα και όπως είπε η κυρία Βερζιά, υπάρχουν θέματα αρχής με το οποίο διαφωνούμε. Το ξέρω, ναι, πράγματι. Υπάρχουν και άλλα πάνω στα οποία μπορούμε να πετύχουμε ευρεία συνένεση. Τώρα για τα θέματα αρχής, τα οποία ανέφερε η κυρία Βερζιά. Μετά τις συναντήσεις με τους σκιώδες εισηγητές βλέπω ότι υπάρχει μια πλειοψηφία στην Επιτροπή μας. Οπότε, αν μπορέσουμε, να συμφωνήσουμε, θα συμφωνήσουμε, αλλιώ θα ακολουθήσουμε τον κανόνα της πλειοψηφία. Αυτό λέει η δημοκρατία. Τι να κάνουμε. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε, Κάρλος. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Δύο μόνο πήρατε το λόγο, αλλά η συζήτηση ήταν ιδιαίτερα επικοδομητική. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Και Μαρή Κριστίν και σαν ευχαριστούμε. Έχουμε άλλο ένα θέμα πριν περάσουμε στην ψηφοφορία. παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της πρώτες Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους τρίτους υπηκόους όταν περνούν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες είναι οι απαιτήσει, οι διατάξεις κλπ. Και δυστυχώς εγώ είμαι ο εισηγητής. Δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στα πλαίσια των προπαρασκευαστικών μέτρων για τον Brexit, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 13 Νοεμβρίου εξέδωσε μία απόφαση προκειμένου να επικαιροποιηθεί ο κανονισμός 539 του 2001, ο οποίος έχει κωδικοποιηθεί και έχει δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, η κωδικοποιημένη μορφή του κανονισμού αυτού. Έχετε λοιπόν πλέον το νέο κανονισμό ο οποίο έχει κωδικοποιημένη μορφή και θα πρέπει να προσέξουμε τώρα και την αντιστοίχηση των διαφορετικών άρθρων που περιλαμβάνονται στη μία και την άλλη εκδοχή. Όλα αυτά γίνονται στα πλαίσια της προετοιμασία για το Brexit. Αν Ξέρετε ότι προβλέπεται εκτό απρόπτου ότι θα αποχωρήσει στι 30 Μαρτίου του 2019 το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα γίνει επομένω τρίτη χώρα. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει με του υπηκόου του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι Βρετανοί πολίτε και οι οποίοι θα θέλουν να διασχίσουν τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να ξέρουμε αν οι υπήκοοι αυτοί θα υπόκεινται σε υποχρέωση θεώρηση ή αν θα παλάσσονται από την υποχρέωση αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει απόλυτη σαφήνεια όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Αν θα πετούνται δηλαδή θεωρήσει για του υπηκόου του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι Βρετανοί πολίτε. Υπάρχουν, όπω ξέρετε, διάφορα κριτήρια στον κανονισμό του Συμβουλίου τον νέο πλέον, τον κωδικοποιημένο 1806, στο άρθρο 1 του νέου αυτού κανονισμού προβλέπει το συγκεκριμένα κριτήριο που λέμε ότι κατά περίπτωση θα πρέπει να εξετάζουμε, να αξιολογούμε την κατάσταση μιας χώρας για να δούμε τελικά αν οι πίκοη της τρίτης αυτής χώρας θα υπόκεινται σε υποχρέωση θεώρησης και αν τελικά θα εισαχθούν στο παράρτημα 1, στο παράρτημα 2. Έχουμε την παράνομη μετανάστευση, τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια, οικονομικά συμφέροντα, το εμπόριο, οι εξωτερικές σχέσεις περιλαμβάνονται στα κριτήρια αυτά, καθώς επίσης και το ζήτημα της αμοιβαιότητας και της περιφερειακής συνεκτικότητας και συνέπειας. Εξετάσαμε λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κριτήρια αυτά σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο και ασχοληθήκαμε επίσης και με τα στοιχεία ασφαλείας των ταξιδιωτικών εγγράφων του Ηνωμένου Βασιλείου και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι υπήκοοι του Μένου Βασιλείου που είναι Βρετανοί πολίτε θα πρέπει να ενταχθούν στο παράρτημα 2 του κανονισμού, δηλαδή θα ανήκουν στου υπηκόου εκείνου, στι χώρε μάλλον εκείνε, οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρηση. Στην ε, αιτιολογική έκθεση ε, Σα δίνουμε περισσότερα στοιχεία. Αναφερόμαστε στο κράτο δικαίου, αναφερόμαστε στην γεωγραφική εγκύτητα, ε, στου οικονομικού δεσμού που έχουμε με το Ηνωμένο Βασίλειο και στις συνθήκες εργασίας που θα ισχύουν στο μέλλον και στις συνθήκες ταξιδίου που θα ισχύουν στο μέλλον μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου ως τρίτη χώρα πλέον και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν έντονοι οικονομικοί δεσμοί, πάρα πολλά ταξίδια τα οποία θα γίνονται για οικονομικούς λόγους αλλά και λόγους αναψυχής και θεωρούμε ότι τα ταξίδια αυτά θα συμβάλλουν στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασιστήκαμε επίσης σε κάποια στατιστικά δεδομένα στον αριθμό των ε, ταξιδιών που γίνονται από τις δύο πλευρές, ε, στις εισαγωγές, στις εξαγωγές, καθώς επίσης και στα χρηματικά ποσά τα οποία δαπανώνται στα πλαίσια των ταξιδιωτικών αυτών. Επίσης, ε, θεωρήσαμε ότι και για το νέο σύστημα αιτίας ε αλλά και για το σύστημα εισόδου-εξόδου θα πρέπει και εκεί πέρα να έχουμε εφαρμογή των συστημάτων αυτών για τους υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι Βρετανοί πολίτες και αυτό ουσιαστικά θα μετριάσει οποιοδήποτε κίνδυνο ενδεχομένω που να υπάρχει σε σχέση με την μετανάστευση και βέβαια θα γίνονται για απαραίτητη έλεγχη σε συγκεκριμένε βάσει δεδομένων όσον αφορά του Βρετανού πολίτε που θα ταξιδεύουν προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νομοθετική λοιπόν πρόταση όσον αφορά τι διατάξει αυτέ περιλαμβάνει τρία νέα άρθρα. Στο άρθρο 1 σημείο 2 γίνεται μια αναφορά στο Μένο Βασιλείο, όπου το Ηνωμένο Βασίλειο θα περιλαμβάνεται πλέον στο παράρτημα 2. Στο σημείο 3 του άρθρου 1 έχουμε του Βρετανούς υπηκόους που δεν είναι Βρετανοί πολίτες, γιατί υπάρχουν, υπάρχουν άλλοι Βρετανοί υπήκοοι οι οποίοι ήδη εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογή του κανονισμού αυτού. Ουσιαστικά η πρόταση θα ισχύει μόνο στους Βρετανούς πολίτες που είναι υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν προκειμένου και που μπορούν ούτως ή άλλως να ταξιδεύουν και θα ταξιδεύουν στο μέλλον προ τι χώρε της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς θεώρηση. Είπαμε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η πρόταση αυτή να επηρεάσει την περιοχή μεταξύ Ιρλανδία και Ηνωμένου Βασιλείου και γίναν και κάποιε τεχνικέ τροποποίησει στον κανονισμό αυτό. Τροποποίηση του άρθρου 4 σημείο 2 Δέλτα, όπου γίνεται διαγραφή τη αναφορά στο Ηνωμένο Βασίλειο γιατί τα όσα λέγονται εκεί αφορούν αυτή τη στιγμή το Ηνωμένο Βασίλειο ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Σέγγεν. Παρ' όλα αυτά, στα πλαίσια της διάταξης αυτής, αλλά σε μία άλλη παράγραφο, την παράγραφο D στο άρθρο 4.2, θα δίνεται η δυνατότητα να απαλλάσσεται το Ηνωμένο Βασίλειο από την υποχρέωση θεώρησης και θα γίνεται ειδική αναφορά στους απάτριδες οι οποίοι δεν έχουν την πικότητα καμίας χώρας και οι οποίοι διαμένουν στην, στο Ηνωμένο Βασίλειο και των οποίων η άδεια διαμονής θα αναγνωρίζεται από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως γίνεται και τώρα. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να ενημερώνει τα υπόλοιπα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με αυτό το άρθρο του κανονισμού. Μια άλλη τεχνική τροποποίηση που γίνεται, η οποία θα επέλθει αυτόματα βέβαια με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πάλι στο άρθρο 4.2α. Τα κράτη-μέλη μπορούν να προβλέπουν συγκεκριμένες διατάξεις όσον αφορά την συμπερίληψη υπηκών του Ηνωμένου Βασιλείου στο παράρτημα 1 του κανονισμού 539. Θα πρέπει και εδώ πέρα πάλι όμως να γίνεται μια κοινοποίηση από τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα της αμοιβαιότητα. έχουμε στο άρθρο 2 συγκεκριμένη αναφορά. Θα γνωρίζετε ενδεχομένω ότι η κυβέρνηση του μέν Βασιλείου είχε πει ότι δεν θα απαιτήσει θεώρηση για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ταξιδεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για διαμονή σύντομης διάρκειας ή για επαγγελματικούς λόγους. Στο άρθρο 2 λοιπόν της πρότασης τονίζουμε περισσότερο το κριτήριο αυτό της αμοιβαιότητος λέγοντας ότι σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο καθιερώσει υποχρέωση θεώρησης για τους υπηκόους τουλάχιστον ενός κράτους μέλους τότε εφαρμόζεται ο, μηχανός, ο μηχανισμός αμοιβαιότητας που προβλέπεται ήδη στον κανονισμό και θα πρέπει τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να εφαρμόσουν το μηχανισμό αμοιβαιότητος αμελητή. Προβλέπεται λοιπόν η άμεση εφαρμογή της, του συστήματος αυτού αν δεν υπάρχει αμοιβαιότητα από πλευράς Ηνωμένου Βασιλείου. Ξέρετε ότι στα πλαίσια του μηχανισμού αμοιβαιότητος προβλέπεται ότι πρώτα θα υπάρχει μια κοινοποίηση από τα κράτη-μέλη. Κράτη-μέλη θα μας λένε δηλαδή ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν σέβεται ε, την αρχή αμοιβαιότητος και εν συνεχεία θα κινητοποιεί το μηχανισμό. Έπειτα στο άρθρο 3 έχουμε τη θέση σε ισχύ. Προβλέπεται ότι ο κανονισμός αυτός θα αρχίσει να ισχύει στις 30 Μαρτίου του 2019, την ημερομηνία τη αποχώρησης δηλαδή του Μανι Βασιλείου. Εφαρμόζεται ο κανονισμός από την επόμενη ημερομηνία κατά την οποία το δίκαιο τη Ένωση πάβει να εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκτό και αν προβλεφθεί στα πλαίσια της Συμφωνίας Αποχώρησης μια άλλη συμφωνία ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ομόφωνα μαζί, μαζί με τον Ηνωμένο Βασίλειο αποφασίσουν μια άλλη ημερομηνία αποχώρησης. Αυτά εν συντομία όσον αφορά την πρόταση αυτή κανονισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά και από το Συμβούλιο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κινηθούν γρήγορα έχοντα κατά νου ότι η πρόταση αυτή κανονισμού θα πρέπει προφανώ να εγκριθεί πριν τι 30 Μαρτίου 2019. Αυτά όσον αφορά το περιεχόμενο τη πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μα ενημερώσατε επώδυνο όλα αυτά που άκουσα. Ενδεχομένω εγώ να το εκλαμβάνω έτσι. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την λεπτομερέστατη αυτή παρουσίαση. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ε, παρατηρήσει από του συναδέλφου. Θα ήθελα βέβαια να έπαινε και μία τροπολογία με την εξαίρεση διεξαγωγής δημοψηφίσματος μέχρι τότε. Τέλος πάντων, το λέω αυτό αστειευόμενος κάπως. Ξέρετε πάντως ότι θα πρέπει να έχουμε και ένα σχέδιο έκθεσης μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου. Μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, ιδίω για το Μένο Βασίλειο, για την πολιτική στον Μένο Βασίλειο. Πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν μέχρι τότε. Πάντω, συνεχίστε εσεί με την επεξεργασία όλων αυτών των διατάξεων για το καθεστώ τη τρίτη χώρα. Δεν πρέπει να τίποτα λιγότερο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν παρατηρήσει από του συναδέλφου. Μέχρι στιγμή δεν έχουμε ούτε καν σκιώδει εισηγητέ. Σα ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πολύ λεπτομεριακή αυτή παρουσίαση που κάνατε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα διακόψουμε πάλι μέχρι τις 5.30. Τότε προβλέπεται η αρχή της ψηφοφορία. Υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι που ακόμα ταξιδεύουν και έχουμε να ψηφίσουμε και σημαντικές εκθέσεις. Θα ήθελα λοιπόν να επιστρέψουμε στις 5 και 20, το λέω αυτό προς τους συντονιστές και σας παρακαλώ πολύ ενημερώστε όλους τους αδέλφους να επιστρέψουν και να έχουν βέβαια και τις κάρτες τους για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Διακόπτουμε μέχρι τις 5 ε, και 20. Um, uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, για τους αναπληρωτές ε, συναδέλφους, να υπενθυμίσω ότι χρειάζεται, χρειάζεται τις ηλεκτρονικές σας κάρτες, οπότε όσοι δεν είναι μαθημένοι και τακτικά μέλη, να σας υπενθυμίσω ότι χρειάζεστε τις ηλεκτρονικές κάρτες. Ε, μπορείτε να τις πάρετε εδώ από τον τρίτο όροφο. Είναι όλες οι ψηφοφορίες ηλεκτρονικές. Οπότε πηγαίνετε πάρτε την ε, καρτούλα σας. Χρειάζεται την κάρτα για να ψηφίσετε. Ειδικά προς ε, τα αναπληρωματικά μέλη. Και 20 ψηφίζουμε. Welcome, colleagues. <clears throat> Uh, we, begin our votes very long. Καλώς ήρθατε συνάδελφοι. Λοιπόν, ξεκινάμε τις ε, ψηφοφορίες, οι οποίες θα είναι μακροσκελέστατες. Λοιπόν, να υπενθυμίσω στους συναδέλφους που δεν είναι τακτικοί εδώ πέρα, ότι οι ψηφοφορίες είναι όλες ηλεκτρονικές, οπότε παρακαλώ να έχετε τις κάρτες σας αν δεν τις έχετε εδώ στον τρίτο όροφο μπορείτε να λάβετε κάρτες ξεκινάμε με την πρώτη ψηφοφορία για την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας για τις ανθρωπιστικές βίζες Χουάν Φερνάντο Λόπεζ Αγγιλάρη είναι Μετά την απόφαση της διάσκεψη των Προέδρων και την απόφαση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, των συντονιστών δηλαδή στι 19 Νοεμβρίου, η Επιτροπή μας ε, αξιοδοτήθηκε να συντάξει ένα ψήφισμα σύμφωνα με το άρθρο 225 της Συνθήκης και το άρθρο 46 των κανονισμών του Κοινοβουλίου. Έχουμε 36 τροπολογίες που έχουν κατατεθεί Δεν ξέρω αν ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ θέλει να μιλήσει. ναι, αλλά να πω ότι και ο κύριος ε, Μπέκερ έχει πει ότι αποσύρει όλες του τις ε, τροπολογίες επί του θέματος. Κύριε Λόπες Αγγιλάρ, έχετε τον λόγο πριν περάσουμε στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σωστά το είπατε. Κράτησε πάρα πολύ η διαδικασία μέχρι να φτάσουμε εδώ και μας μένει και πολλής δρόμος στην ψηφοφορία ακόμα. Δουλέψαμε σκληρά. Ιδιαίτερα τις τελευταίες αυτές εβδομάδες, τελευταίες ε, μέρες, τελευταίες ώρες. Γι' αυτό και θέλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους που είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν την προσπάθεια που έγινε για να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς. Να ξέρετε ότι ο κατάλογος ψηφοφορίας έχει δουλευτεί πολύ Προσπαθήσαμε να πετύχουμε μια ισορροπία και καταφέραμε να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ θέσεων που ήταν αρκετά αντιδιαμετρικές μεταξύ τους στην αρχή. Αλλά πιστεύω ότι καταφέραμε να πετύχουμε συμβαστικές προτάσεις αποδεκτές από όλους. Και έτσι τώρα έχουμε την ευκαιρία να πετύχουμε να ενσωματωθεί ο κώδικας αυτός έγκαιρα, τον παρουσιάζουμε για να σωματωθεί ακριβώς και από την άλλη μεριά έχουμε και τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις ως έκθεση πρωτοβουλίας. Για έναν καλό σκοπό για αυτούς που τόσο πολύ το χρειάζονται. Αυτοί που κινδύνεψαν στη Μεσόγειο για να μπορέσουν να βρεθούν στην ε, Ευρώπη ή για αυτούς που έχασαν και τη ζωή τους, γιατί ξέρετε ότι δεν έχουν νόμιμο τρόπο να το πετύχουν αυτό. Οπότε με αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα ψηφίσουμε σήμερα θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και ευχαριστώ πολύ τους και όδες εισηγητές, όλους που έβαλαν τα δυνατά τους με τις δικές τους προϋποθέσεις, αλλά όσοι υπερψηφίσουν τους ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Χουάν, και τους ε, σκιώδεις συζητητές. Περνάμε στην ψηφοφορία. 16, 17, 18 και 32 όλες μαζί άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτονται. 20 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 25 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 27 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 28 ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Η 29 ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 30 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 31 έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ναι, απορρίπτεται. Ε, Τη αναφορά 1 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 2 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Εκτιμώντας ε, τροπολογία 3 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 6 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 7 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Καλώς. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, όλες μαζί άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. απορρίπτονται. Ευχαριστούμε, Μπίργκιτ. Το παράρτημα μπορούμε να το κάνουμε όλο μαζί. Όχι. Λοιπόν, 33 άρχεται η ψηφοφορία. Συγγνώμη, εκεί πέρα χάρηκα. Πέρας. Απορρίπτεται. 34 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 35 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Να Και 36 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται και η τελική ψηφοφορία με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή. 37 υπέρ 10 κατά 3 αποχές συγχαρητήρια περνάμε τώρα στην επόμενη ψυχοφορία να σας ε, προειδοποιήσω εδώ πέρα δεν είχαμε πολλές συμβαστικές ε, τροπολογίες λοιπόν ψηφίζουμε για τον κώδικα Βίζεσια για να πάμε σε διαπραγματεύσεις και για τη σύνθεση διαπραγματευτικής ομάδας και πάλι ο Χουάν Φερνάντο Λόπες Αγγιλάρα. Έχουμε συμφωνήσει στις ομβαστικές τροπολογίε, αλλά επειδή δεν υπήρχε αρκετό χρόνος έχουμε πολλές μεμονωμένες τροπολογίες. Ε, δηλαδή θα τραβήξει πολύ. 95 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 96 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 5 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Συνάδελφοι. Είναι κάποιος παραπάνω από το ΕΛΚΑ. Ρομπέρτο. Εντάξει, λύθηκε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τραν 39. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 97. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 98. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 99. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας απορρίπτεται 103 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 100 και 101 ταυτόσιμες άρχεται η ψηφοφορία πέρας δεκτή 102 άρχεται ψηφοφορία Πέρας. Απορρίπτεται 104 για τη Πέρας. Απορρίπτεται. 105 άρχεται η Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 6 αρχή ψηφοφορία. Πέρας. Ε, όχι, είχε τελειώσει αυτό. Δεκτό. Τροπολογία 7 αρχή της ψηφοφορία. Δεκτή. Τροπολογία 108 αρχιτή ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 109 αρχιτή ψηφοφορία. Πέρας. Τροπολογία 8. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 110 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 9 και 112 ταυτόσημες άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 111. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 114. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 115. Άρχεται η ψηφοφορία. ημέρας. Δεκτή. Θέλετε να τις κάνουμε όλες μαζί. Ναι. 116 ε, με 121. Για να δούμε. Άρχεται Όχι. Όχι δεν μπορούμε. Όχι, Μπίργκιτ, όχι, όχι. Λοιπόν, ε, τώρα να. Σπαταλήσαμε χρόνο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 116 λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Ε, θα πάω σου ευρώ 117 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 119 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 120 αρχές ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 11 αρχιετή ψηφοφορία. Εκατόν αρχιετή ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τι θέλετε. 122 αρχή ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 123 αρχή ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 124 άρχη ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 126 άρχη ψηφοφορία πέρας Απορρίφθηκε. 125 άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. 127 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τραν 49 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 128 άρχιτη ψηφοφορία. απορρίπτεται. 129 έρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Ξανά άρχισε άλλο Μαρτί γίνεται. Απορρίπτεται. Τραν 42. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τραν 46. Άρχεται ψηφοφορία. Κάτι ξεχάσαμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 130 έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 131 έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 132 έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Πέρας. 133 με ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησε το ΕΛΚΑ για τη ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίφτεται. 134 αρχιετή ψηφοφορία και η 12. Με ονομαστική ψηφοφορία ζήτησε το ΕΛΚ. Ναι. Συγγνώμη, δεν είναι 134 και 12, άκυρο. 135 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και απορρίπτεται. Συμβαστική 3 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τώρα πάμε στην τροπολογία 4, συμβαστική 4, στη σελίδα 10, άρχεται η ψηφοφορία. Συμβιβαστική 4. Πέρας. Δεκτή. 159 ψηφοφορία. Σελίδα 13 στο δικό μου το χαρτί. Συγγνώμη, ναι. Ε, πρέπει να τα λέω αυτά. Πέρας. Απορρίπτεται. Τραν 5. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 160 και τραν 55 ταυτόσημες. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτονται. Συμβαστική 5 άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Πάμε συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 6, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 168, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 169, με συγχωρείτε, τροπολογία 27, διορθώνει ο πρόεδρος. Ναι, ναι, το είπα σωστά τώρα, τροπολογία 27. Σας δοκιμάζω να δω αν παρακολουθείτε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 169. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 170. Ψηφίζουμε. Πέρας. Και απορρίπτεται. Τροπολογία 174. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 175, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 176, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 177 και 178 ταυτόσιμες άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτονται 179. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τραν συμβαστική υπαριθμών 2. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 180. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 181. Άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 29. Άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 182. Άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 130, 184, 185 και 365 και 31 μαζί είναι ταυτόσιμες. Άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνονται. Περνάμε στην 31, άρτη ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Τροπολογία 186, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Συμβαστική 7, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 195 και 196 μαζί με ονομαστική κλίση μετά από αίτημα του ΕΛΚ, άρθρη ψηφοφορία. Πρέπει να διαβάσω το κείμενο εδώ. 195 και 106 από κοινού ονομαστική κλίση μετά από αίτημα του ΕΛΚ πέρας. Όχι ακόμα. Είστε πολύ αργοί. Τι συμβαίνει. Ψηφίσατε όλοι πέρα. Απορρίπτεται. Απορρίπτονται, μάλιστα. 34. Άρθρο ψηφοφορία. Πέρα. Απορρίπτεται. Τροπολογία 197. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. 198. Όχι. 100. Περνάμε στη 201, άρτη ψηφοφορία, με ονομαστική κλίση μετά από αίτημα του ΕΛΚ. Πρέπει να το διαβάζω αυτό που ό,τι μου λένε. Πέρας. Εγκρίνεται. 203, τρία. ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 204. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβασική τροπολογία 8. Άρχιτη ψηφοφορία. Με ονομαστική κλίση μετά από αίτημα του ΕΛΚ. Τι να πω, πρέπει να το διαβάσω από ό,τι μου λένε. Λοιπόν, πέρας. Εγκρίνεται. 225. 225 άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 226 άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 227 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 228 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 230 τώρα άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 38 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 231 άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 233 άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 39 άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 234 άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 235 άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 236 άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 237 άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 238 άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στη 239, 240 και 241 ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε από κοινού άρτη ψηφοφορία. Πέρας. απορρίπτονται. «242 άρτη ψηφοφορία». Πέρας. Απορρίπτεται. 243 άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 41. Άρτη ψοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τρανθρωπολογία 74. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τραν 75. Άρτη ψηφοφορία. Πέρες. Εγκρίνεται. Τραν 76. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 244 άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 245 άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 242 άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. 247 άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 43 άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 249 άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 44. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 250. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 251. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 252 άρτη ψηφοφορία. Πέρας. 257 άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 253 άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 254. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 255. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 256. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 258. άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 259 άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 260 άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 261 άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 262. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται 264. Άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 265. Άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 266 με ονομαστική κλίση μετά από αίτημα του ΕΛΚ, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογίες 45 και 267 που είναι ταυτόσιμες με ονομαστική κλίση μετά από αίτημα του ΕΛΚ, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτονται. Τροπολογία 268. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 269. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 270. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 271 άρχιτη ψηφοφορία πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 273 άρχιτη ψηφοφορία πέρασε. Απορρίπτεται. 274 άρχιτη ψηφοφορία πέρασε. Εγκρίνεται. 275. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 276. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 47 και 277 μαζί είναι ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε. Πέρας. εγκρίνονται. 278 άρτη ψηφοφορία. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος. Ψηφίζουμε την 279. Άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 280 άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 281 άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 282 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται 284. Άρτη ψηφοφορία πέρασε. Εγκρίνεται. Περνάμε στις λογικές σκέψεις, τροπολογία 49 με ονομαστική κλίση, μετά από αίτημα του ΕΛΚΑ, ψηφίζουμε. Πέρασε. Και εγκρίνεται. 50, σας το συγγνώμη, όχι την 51, λέει ο πρόεδρος, όχι, όχι, την 52 ψηφίζουμε. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τροπολογία 52, μονομαστική κλίση μετά από έτοιμα του ΕΛΚΑ. Άρχεται ψηφοφορία. Σα ζητώ συγγνώμη, αλλά πρέπει να διαβάσω την υποσημείωση εδώ. Πέρασε. Και απορρίπτεται. Περνάμε τροπολογία 53. Άρχτη ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται τροπολογία 54, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Και απορρίπτεται. Τροπολογία παριθμών 1, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 55, ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται 56 άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 58 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 59 άρτη ψηφοφορία. Ψηφίσουμε την 59. Για την Κατερίνα το λέω αυτό. Πέρας. Και απορρίπτεται. Τραν συμβαστική υπαριθμών 3, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. Τροπολογία 60, άρχιτη ψηφοφορία. Σας ζητώ συγγνώμη που έδινε υποδείξει ένα μέλο των σοσιαλιστών. Λοιπόν, ψηφίζουμε την 60, πέρας και εγκρίνεται. Τροπολογία 61, άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 62, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Κοντεύουμε. Φτάνουμε στο τέλος. Λοιπόν, σας το συγγνώμη, ταυτόσημη ήταν για την προηγούμενη. Επομένως πάμε στην 65, λέει ο Πρόεδρος. Σας το συγγνώμη, έχω αρχίσει να κουράζομαι, λέει ο Πρόεδρος. Ψηφίζουμε την 65. Πέρας. Και απορρίπτεται. Πάμε στην τροπολογία 66, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τράνε υπαριθμών 17 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τραν 18 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 67 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Τροπολογία 68, ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 69, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 70, Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 71. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τράνη παριθμόν 20. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 73 με ονομαστική κλίση μετά από έτοιμα του ΕΛΚ. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. Όχι, σε ζητώ συγγνώμη. Τι συνέβη ακριβώς, λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, ψηφίσουμε ακόμα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεν ξέρω τι συνέβη, αγαπητοί συνάδελφοι, το συγχνώμη. Περνάμε στην τροπολογία 74. Διορθώνει πρόεδρος, τροπολογία 76, άρτη ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 76. Πέρασε. Απορρίπτεται. Ψηφίσουμε μαζί τις 3, 77 και 78, άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτονται. Τροπολογία 79. Άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 80, μάλλον 81. Άρτη ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 81. Πέρασε. Απορρίπτεται 82. Άρτη ψηφοφορία. Ψηφίζουμε το 82. Πέρας. Εγκρίνεται. Οι επόμενες δύο, 26 και 27 από την Τραν, δεν εγκρίθηκαν στην Επιτροπή Τραν, επομένως δεν πρόκειται να τις ψηφίσουμε. Περνάμε έτσι στην 83, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 84, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται τροπολογία 86. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 87. Μονομαστική κλίση μετά από αίτημα του ΕΛΚ. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 88, άρχιτη ψηφοφορία. Με ονομαστική κλίση. Με τα αποέτοιμα του ΕΛΚ. Όλος περιέργος. Πέρας. Απορρίπτεται. 89. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας απορρίπτεται. Τροπολογία 90, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 91, ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τραν, τροπολογία 33, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. Τροπολογία 92, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τραν συμβαστική τροπολογία 4, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 93. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 94. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. Τώρα ψηφίσουμε το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική κλίση άρρηκτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας και γκρίνεται 27 υπέρ 15 κατά 4 αποχές. Και τώρα ψηφίζουμε την απόφαση έναρξης διεργανικών διαπραγματεύσεων, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 28 υπέρ, 13 κατά και 4 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Συγχαρητήρια σε όλους τους σκιώδεις εισηγητές και σε όλο το προσωπικό. Sorry. So we're short of the absolute majority by one. Οπότε δεν έχουμε απόλυτη ψηφοφορία, μας λείπει, απόλυτη πλειοψηφία μας λείπει ένας. Όπως βλέπετε έχουμε την απόλυτη πλειοψηφία με δύο ψήφους. Δεν έχουμε την απόλυτη πλειοψηφία, μας λείπουν δύο ψήφοι. Σας ευχαριστώ όλους για τη βοήθειά σας. προστασία του ευρωπαϊκού προπολογισμού σε περίπτωση γενικευμένων αδυναμιών όσον αφορά το κράτος δικαίου στις χώρε μέλη. Η συγγητής μας είναι ο κύριος Τερικάμπρα. Μήπω θέλετε το λόγο πριν αρχίσουμε, παρακαλώ. Ναι, θέλω να διευκρινίσω τι υποστηρίζουμε, να επεκτηθεί το πεδίο εφαρμογή της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να υπάρχει μία ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα βοηθάει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αξιολόγηση, να ενημερωνόμαστε για τα ευρήματα του πάνελ αυτού και να ενισχύσουμε τους δεσμούς με τις αρχές του προπολογισμού. Τη μνήμα στο άρθρο 7 την αφήνουμε με το πνεύμα συμβιβασμού και επίσης αφήνουμε και την μνήμα στη δημοκρατία τι περιμένουμε τώρα από την ψηφοφορία. Στήριξη στη γνωμοδότηση, η οποία είναι περισσότερο φιλόδοξη από την πρόταση τη Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών. Και ελπίζουμε οι πολιτικέ ομάδε να στηρίξουν την πρόταση αυτή και στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Τέρη Κάμπρα. Ψηφίζουμε τροπολογίες 27 και 28 που είναι ήδη μαζί. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβαστική τροπολογία 4. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 136. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί όλες αυτές τις τροπολογίες. Ναι. 136 με 151. Όχι, ωραία. 136. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίπτεται. 137. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίπτεται. 138. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. 139. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίπτεται. 141. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίπτεται. 142. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίπτεται. 143. Ψηφίστε. Α, όχι, όχι. 144 ψηφίζουν. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίπτεται. 145. Ψηφίστε. ήταν 145. Τέλος της ψηφοφορίας απορρίφθηκε. 147. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίπτεται. 149. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίπτεται. 151. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Απορρίπτεται 152. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίπτεται 153. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίφθηκε 155-156 ψηφίστε. Τέλος. Απορρίπτονται. 160 ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίπτεται. 161 ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. 162. 162 ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. 163. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. Συγγνώμη, Μπάρμπαρα, λέει ο πρόεδρος. 164 ψηφίστε. Τέλος. Απορρίπτεται. 165. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίπτεται. 167. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίπτεται. Κάνω ό,τι μπορώ, Μπάρμπαρα, αλλά οι συντονιστές δεν βλέπω. 169. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. 170. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε και αυτή. Τροπολογία 32. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια Μπάρβαρα. 33. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Εγκρίθηκε και αυτή. Αιτιολογικές σκέψη. Συμβαστική 6. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία Τώρα, τελευταία σελίδα. Τροπολογία 80. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε 81. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίπτεται. 91. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίπτεται. 92. Τέλος. Απορρίπτεται. 83. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίπτεται. 84. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίπτεται. 85. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. 86. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίφθηκε. 87. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίφθηκε. 90. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίφθηκε. 89. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. Τελική ψηφοφορία ονομαστικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε 33 ψήφοι υπέρ, 10 κατά, 3 αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Τερικάμπρας. Τώρα περνάμε σε άλλη μία έκθεση του κύριου Τερικάμπρας. Πρόκειται για την κατάσταση θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Τερικάμπρας, να ψηφίσουμε ή θέλετε να πείτε κάτι πριν. Ναι, κάτι έχω να πω, αλλά αργότερα γιατί είμαστε όλοι κουρασμένοι. Ας ψηφίσουμε. Ψηφίστε υπέρ παρακαλώ. Ωραία. Ωραία ομιλία. Σας ευχαριστώ πάντως, λέει ο Πρόεδρος, έτσι καλλιώς όλους που είσαστε τόσο καλοί με την ψηφοφορία. Κανένας δεν μου γκρινιάζει. Ευχαριστώ για την πειθαρχία. Λοιπόν, αρχίζουμε τροπολογία 86. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία αριθμός 1. Ψηφίστε παρακαλώ. Έκανε λάθο. Α, συγγνώμη, συγγνώμη λέει ο Πρόεδρος. Συγγνώμη. Προσπαθώ ναι, να τελειώσω γρήγορα. Βασικά. Συγγνώμη, 86 ήταν, οπότε τώρα είναι 87 βέβαια. Ψηφίζουμε την 87. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίπτεται. 89. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίπτεται. 90. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. 93. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. 94. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίφθηκε. 95. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίπτεται. 96. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Απορρίπτεται. 97. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίφθηκε. 98. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. Συμβαστική αριθμός 1. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική τροπολογία 1α. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβαστική τροπολογία 4α για τα δικαιώματα των παιδιών. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβαστική τροπολογία... Α, συγγνώμη, διορθώνω ο Τροπολογία 147 πρώτα. 147. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβαστική τροπολογία 2. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβαστική τροπολογία 4B. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 52. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική πολιτική. Τρία λέει ο πρόεδρο. αλλά όχι, μετά την 52 έχουμε την 145. 145. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίπτεται. 185. 185 με 190 μαζί να τις ψηφίσουμε. Εντάξει, ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν. Ψηφίστε παρακαλώ. Ναι, ναι, θα το κάνουμε πιο συχνά. Ωραία. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκαν. 192 με 194 μαζί ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίφθηκαν. Συμβαστική 3. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 4. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Μπράβο κύριε Τερικά, προσκαλέ αυτές τι συμβαστικές. 265 τώρα. Μπορείτε να ψηφίσετε. 265 τροπολογία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίθηκε. 269. Ψηφίστε. Τέλος. εγκρίθηκε. Συμβαστική τροπολογία 6α. Ψηφίστε. Για το Brexit, ναι, είναι καταθλιπτικό. Τι σημαίνει, όχι Brexit, καλά. Τι να κάνουμε, ψηφίσαμε να κυρωθεί το Brexit, λοιπόν. Τέλος της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Ακυρώνεται το Brexit, λέει ο πρόεδρος αστευόμενο. Συμβαστική τροπολογία 5 ψηφίστε. Τέλο Εγκρίθηκε. Συμβαστική 6. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Καλή και αυτή. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 312. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίπτεται. 313. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6B. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 7. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Ωραία. Τροπολογία 381. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της προφορίας. Απορρίφθηκε. Τώρα πάμε. Τροπολογία 408. Ψηφίστε παρακαλώ. Δεν μπορούμε όλες μαζί, μία-μία θα τις ψηφίσουμε αυτές. Τέλος απορρίφθηκε. 409 ψηφίστε. Τέλος. Απορρίπτεται. 410 ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. 411 ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. 412. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. 413. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίπτεται. 414. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίνεται. 415. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίπτεται. 4-16 Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Ετουλικές αναφορές. Η συμβαστική 7α. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. Αιτιολογικές ε, σκέψεις. Συμβαστική 8. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 22. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίπτεται. 24. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίπτεται. Συμβαστική 9. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική 12. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίνεται. 79. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 80. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίφθηκε. Τελική ψηφοφορία τώρα, με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι, τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε 31 ψήφοι υπέρ, 13 κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια κύριε Τερικάβρας και πάλι. Οπότε, συνάδελφοι, είναι προτελευταία, όχι, η τρίτη από το τέλος. Λοιπόν, συνεχίζουμε όπως και να έχει. Σας ευχαριστώ. Θα μια χαρά. Και σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Είστε έτοιμοι. Πάμε κατευθείαν στην τροπολογία 11. Πάμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Αν θέλετε διάλειμμα, πείτε το. Όχι, όχι. Ναι, έτσι. Εγώ χρειάζομαι διάλειμμα, αλλά τέλος πάντων. Πέρασε. Δεκτή 12, άρχεται η ψηφοφορία. Ναι, ναι, έχετε δίκιο, γιατί άμα γίνει διάλειμμα δεν θα επιστρέψουμε. Πέρας. Δεκτή 13 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 14 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 15 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Εκτιμώντας ένα. Όχι, όχι. Τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτή. 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεκτή. Ε, πέρασε, με συγχωρείτε. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία με ονομαστική ψηφοφορία. αρχιτεκτή. Πέρασε. Να πω ότι δεν σας είπα ποια ήταν η ψηφοφορία. Ζητώ συγγνώμη από την κυρία Γκάλ. Ήταν η έκθεση για ένα ταξιδιωτικό έγγραφο ανάγκης. Ε, ζητώ συγγνώμη, πρώτη φορά εδώ και πέντε χρόνια έχω κάνει κάτι τόσο βλακώδες. Δεν είπα καν τι ψηφίζαμε. Δηλαδή μπορούσαμε να ψηφίσουμε το οτιδήποτε. Θέλετε τον λόγο? Όχι. Συγγνώμη, Κίνγκα. Ωραία. Έχει γίνει τελευταία ψηφοφορία. Ωραία, οπότε ευτυχώ, πέρασε 41 ε, ψήφοι υπέρ 4 κατά. Λοιπόν, σα είπα το θέμα, Ωραία η έκθεση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Λοιπόν, τώρα θα τα πω σωστά. Επαναδέσμευση των υπολείπων ποσών για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου ή σε άλλες δράσεις υπό τα εθνικά προγράμματα. Η συγκεκριά είναι η ειναι Νταλή. Θέλετε να μας πείτε κάτι είναι η προσωρινή συμφωνία που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις Μύρια. Όχι. Ψηφίζει σε άλλη επιτροπή. Α, εντάξει, με κάνετε έτσι. Ρώτησα αν είναι εδώ. Λοιπόν, μία είναι η ψηφοφορία. Άρχεται. Τώρα στα κακοί. Πέρασε. δεκτή. 25, 18 και μία αποχή. Συγχαρητήρια στη Μύρια μου όπου και αν είναι. Μάλλον θα ψηφίζει στην Επιτροπή Μεταφορών. Ευχαριστώ. Το επόμενο είναι ψήφισμα για την επάρκεια της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που παρέχει η Ιαπωνία. Περνάμε στη ψηφοφορία. Τροπολογία 22 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτή. 25 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Πέρας. Απορρίπτεται. 26 άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. 27 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Λοιπόν, 28 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 29. Όχι. 31 άρχεται ψηφοφορία. Αυτό λοιπόν. 31, 32, 33 άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτές. 35 άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 39 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφτεται. Σαράντα. Σαράντα. Πέρας. Δεκτή. Σαράντα τη Άρχιτη Φυσοφορία. Πέρας απορρίπτεται 43 άρχεται η ψηφοφορία πέρας δεκτή 44 που είναι προσθήκη τη 44 λοιπόν ως προσθήκη αλλά σημειώνει ότι αυτό αφορά πολύ περιορισμένες καταστάσεις ω προσθήκη 43. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεκτή. 45 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 46 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απόρριπτεται 47. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 48 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 49 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 50 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απόρριπτεται. 52 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 51 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 53 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 54 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 55 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 56 έρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 57-58 ταυτόσημες έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 59 έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 60 άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. 62 άρχεται. Πέρασε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 61 άρχεται η ψηφοφορία. δεκτή 64 άρχεται το φοβερό είναι αυτό το πράγμα πέρασε δεκτή 65 ως προστίκη άρχεται η ψηφοφορία πέρασε Απορρίπτεται. 69 άρχεται η ψηφοφορία. Α, 69 μάλιστα. Πέρασε. Απορρίπτεται. 68 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 70 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται 71 άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται 72, άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται 73, άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται 74, άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται 75 άρχεται η ψηφοφορία πέρας δεκτή 1 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ε, τροπολογία 2 άρχεται η ψηφοφορία πέρας δεκτή Τέσσερα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται Τρία. έρχεται, Πέρας. Δεκτή. Πέντε. Όχι. Έξι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Α, απορρίπτεται. 8. Έρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 7. Έρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. απορρίπτεται 10 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 9 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 12 άρχεται πέρας απορρίπτεται 13 άρχεται πέρας απορρίπτεται 15 άρχεται πέρας δεκτή 16 άρχεται πέρας δεκτή 17 αρχιετή ψηφοφορία πέρας Απολύπτεται. 17, 18 όχι 18 και 19 ταυτόσιμες πέρας δεκτή 20 αρχιετή ψηφοφορία πέρας Δεκτή. Τελική ψηφοφορία. Ονομαστική. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Τι 28 ψήφιπε, 9 κατά και 7 αποχές. Ω, Παναγία μου, τι γίνεται. Λοιπόν, Ας περάσουμε τώρα στην επόμενη ψηφοφορία. Νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη ψηφοφορία χρονικά που έχουμε κάνει ποτέ. Αλλά κοντεύουμε να τελειώσουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, πάμε στην επόμενη έκθεση «Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». Έγκριση της, του σχεδίου γνωμοδότησης που είχε συντάξει η Σοφίντ Βέλτη η οποία δεν θέλει να πάρει το λόγο, άρα ψηφίζουμε κατευθείαν τροπολογία 13, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3, άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Ως προσθήκη, άρτη ψηφοφορία, πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία πάλι 14, το δεύτερο τμήμα τώρα, το ψηφίζουμε πάλι και αυτός προσθήκη, άρχεται ψηφοφορία, πέρασε. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα τώρα της τροπολογίας 14, άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 16, άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στο λογικέ σκέψεις. Τροπολογία παριθμών 1. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα μονομαστική κλίση, άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 39 υπέρ 2 κατά και μία αποχή συγχαρητήρια στην συντάκτρα νομοδότησης. Λοιπόν, περνάμε τώρα στην πρώτη τελευταία ψηφοφορία θα προσπαθήσω να προχωρήσω γρήγορα. Ενίσχυση τη ασφάλεια των δελτίων ταυτότητα των πολιτών τη Ένωση και των εγγράφων διαμονή που εκδίδονται για του πολίτε τη Ένωση και τα μέλη τη οικογένειά του που το δικαίωμά του στην ελεύθερη κυκλοφορία. Η συγκεκριτή είναι ο κύριο Ντεπρέ Ζεράρ. Θέλει να πάρει το λόγο πριν την ψηφοφορία. Όχι. Άρα ξεκινάμε κατευθείαν ψηφοφορία. Όλοι έχουμε εργαστεί σκληρά για τις εκθέσεις αυτές, άρα ψηφίζουμε αμέσως τροπολογία 69, άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 70, άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 27 άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία παριθμών 1 άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2 άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία παριθμών 3, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Άρτη ψοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε έτσι γρήγορα στη συμβαστική τροπολογία 5. Σε ευχαριστώ Ζεγάχ όχι για την έκθεση στο σύνολό τη, αλλά για τον τρόπο που διεξάγεται η ψηφοφορία με τι συμβαστικέ τροπολογίε που κατέθεσε. Λοιπόν, συμβαστική τροπολογία 5, ψηφίζουμε, πέρα και εγκρίνεται. Περνάμε έτσι, συμβαστική τροπολογία 6, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 8, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. Συμβασική τροπολογία 9. Άρκτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβασική τροπολογία 10. Άρκτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Σημαντική τροπολογία 11. Ψηφίζουμε. Α, πάντα υπάρχει μια μικρή παγίδα, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ψηφίζουμε την 188. Το έκανα για να δω αν έχετε αποκοιμηθεί. Λοιπόν, ψηφίζουμε την 188. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την 189, άρχιτη ψηφοφορία. Ξεχάστηκα και εγώ, λέει ο πρόεδρος. Πέρασε. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 11, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 12. Ψηφίζουμε την συμβαστική τροπολογία 12. Με κάνει και χάνει αυτοποίθησή μου. Λοιπόν, ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία 12. Πέρασε. Εγκρίνεται. Περνάμε στις... Μάλλον, 205 ψηφίζουμε, λέει ο Πρόεδρος. Δεν έχετε αποκοιμηθεί από ό,τι βλέπω. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 71 σε σκέψεις. Άρθρη ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 79. Άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 96 τώρα. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 103. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται 102 άρτη ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 104 άρχεται ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται τροπολογία 106 ψηφίζουμε Τέλος, απορρίπτεται τροπολογία 25, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τροπολογία 26, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελική τώρα ψηφοφορία για το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική κλίση άρθρη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται 32 υπέρ 7 κατά και 3 αποχές. Συγχαρητήρια. Ψηφίζουμε τώρα την απόφαση άνεραξης διοργανικών διαπραγματεύσεων. Άρτη ψηφοφορία παρακαλώ. Ψηφίζουμε την απόφαση άνεραξης διαπραγματεύσεων. Χρειαζόμαστε απόλυτη πλειοψηφία, αγαπητοί συνάδελφοι. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. 35 υπέρ, 7 κατά. Καμία αποχή. Συγχαρητήρια στον εισηγητή, τον κύριο Ντεπχέ. Πολύ ωραία. Περνάμε έτσι στην τελευταία μας ψηφοφορία για σήμερα. Ευχαριστήσω πραγματικά ειλικρινά όλους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 Ψηφίζουμε την τροπολογία 39 άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Ένα άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Περνάμε λοιπόν στην 107. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 109. Και οι 20 της έχουν ταυτόσημες. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας τα συμβαστικη Συμβαστική άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 1-1-5 Άρχητη ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 17 και έκον 21 έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 119. Άρχεται η ψηφοφορία. 118 αποσύρεται. 119. Πέρας. Απορρίπτεται. 120 και 122 αρχή της ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτή. Εκον 23. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Συμβαστική 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 126 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 128. Συγγνώμη, τι μου ξέφυγε. Συγγνώμη, συνάδελφοι. 127 και έκον 25 συγγνώμη ναι άρχεται ναι ναι πέρας δεκτή 128 και ε, όχι 128 μόνο Πέρασε. Ε, σχεδόν φτάσαμε. Λοιπόν, πέρας. Δεκτή. 129 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 131. Α, 27 της έκονα άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 130 αρχιτή ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 131, 32 και 28 της έκονα αρχιτή ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 133 άρχεται πέρας απέριφθητε έκον 29 άρχεται πέρας δηλαδή 134 άρχεται πέρας δεκτή 136 άρχεται πέρασε δεκτή σταματήστε λοιπόν 137 άρχεται δεκτή 138 άρχεται η ψηφοφορία πέρασε Δεκτή. Τροπολογία 4. Συμβαστική άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 5. Συμβαστική άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική 6. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή.

Πέρας. Δίκτυ 22 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 175 άρχεται. Πέρας. δεκτή 176 έρχεται πέρασε δεκτή 177 έρχεται όχι 77 με συγχωρείτε πέρασε δεκτή 177 έρχεται ναι, ναι. 77 ήταν πριν. Την 77 είπα. Ε, τα άκουγε κυρία Χολμαϊρ, είπα 77 και τώρα είμαστε 177. Δεν είπα, είπα η κυρία Χολμαϊρ το άκουσε. Την 77 ψηφίσατε. Θέλετε να την ξαναψηφίσουμε. Ωραία. 177 άρχεται. Ψηφίζουμε. Ωραία. 77. Δεν ξέρω τι συμβαίνει εδώ δηλαδή. Και θα καταψηφίσω αυτή τη φορά. Θα καταψηφίσω. Πέρας, κάπου εδώ σας ε, αποχαιρετούν και οι διερμηνείς, καθώς έχουμε υπερβεί το ωραριό μας. 7 Okay. And the vote is closed. That's carried. Right, Econ 38, open. Four. Closed.